Καλησπέρα σα. Θα... Σήμερα το πρωί στην ε, συνεδρίαση των συντονιστών ελήφθησαν οι ακόλουθε αποφάσει. Εγκρίθηκε το σχέδιο ημερήσια διάταξη τη συνεδρίασης ε, τη Επιτροπή Αναφορών για τις 19 και 20 Φεβρουαρίου του 2020 και οι αναφορές 865 το 2018, 143 το 2019, το 811 2019 θα συμπεριληφθούν. Οι 115 56, 1.40 το 2019 και ε, 10-59 το 2019 θα πάνε με την κατεπίγουσα διαδικασία και θα συμπεριληφθούν στην εμερήσια διάταξη του Φεβρουαρίου. Η ετήσια έκθεση του 2019 για την Επιτροπή Αναφορών δόθηκε στο ICR. E οι συντονιστές συμφώνησαν να ζητήσουν την άδεια να συντάξουν έκθεση για την προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βάσει της ε, Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, ε, βάσει των θεμάτων που την αφορούν και δόθηκε στο ε, στο ΕΛΚ. Επίσης, αποφασίστηκε μια έκθεση για την ε, Τουρκία, για ε, γνωμοδότηση επίσης για την ΑΦΕΤ και την ΙΤΑ, για τις διαπραγματεύσεις και τις μελλοντικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η γνωμοδότηση δόθηκε στο ΕΛΚ. Οι συντονιστές αποφάσισαν ότι η Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να κάνει τις ακόλουθες αποστολές για το δεύτερο εξάμεινο του 2020. Μία αποστολή σε ένα γερμανικό γραφείο ε, πρόνοια των νέων στο Γιούγκενταμ και επίσης ε, μία επίσκεψη στην Ισπανία και επίσης αποφασίστηκε να δοθεί άδεια, να ζητηθεί άδεια να γίνει μία διερευνητική αποστολή στις Ηνωμένε Πολιτείε για να συναντηθούμε με μέλη του Κογκρέσου και να συζητήσουμε τον αντίκτυπο ε, του συμφώνου για τη φορολογική συμμόρφωση των ξένων λογαριασμών. Επίσης, σημειώσαμε τα ονόματα των μελών που συμμετέχουν στην αποστολή στην Βουλγαρία. Επίσης εγκρίθηκε το σχέδιο προγράμματος το κοινή ακρόαση ε, με, μεταφορών και αναφορών για τον τομέα της αεροπορίας και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Ε, θα γίνει ε, θα πρέπει να ζητήσουμε στοιχεία μέχρι 30 Ιανουαρίου. Επίσης αποφασίστηκαν να συζητηθούν οι ακρονάσει και τα εργαστήρια για την επόμενη συναντήρια των συντονιστών. Ζητήθηκε να υπάρξει προπαρασκευαστική μελάτη για την ακρό, ε, ακρόαση για την επιτυχή διαδικασία πρωτοβουλίας των πολιτών και επίσης σημειώσαν την επιστολή της ε, ε Επιτροπής ε, του και αποφασίστηκε να μην γνωμοδοτήσουμε για τον ετήσιο προπολογισμό του 2021. Επίσης, συμφωνήσαμε να υποβάλουμε την πρόταση του Ρινιού για την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την καταπολέμηση της ένδυας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρόταση της ΓΟΕ για την πρόνοια των ζώων για τις μεταφορές, κατά τη μεταφορά. Συγγνώμη. Ο συμβολή στο πρόγραμμα του 2021 και Όσον αφορά τις αμφισβητούμενες συστάσεις, εγκρίθηκαν με τη μορφή που πρότεινε η Προεδρία για τις αναφορές 631, 633, 738 και 780 ε, του 2019. Εγκρίθηκαν όπως πρότειναν οι πράσινοι οι αναφορές 768, 778, 779 και 790 και 782 του 2019 όπως το πρότειναν οι πράσινοι. Όσον αφορά τώρα τα θέματα Β, αποφασίστηκε να μείνουν ανοιχτέ οι αναφορές και να ζητήσουμε περαιτέρω αναφορέ, ε, δράση για την 389, 830, 1146, 665 του 2019 και 65 216 και 310 του 2019. Επίσης συμφωνήθηκε να κλείσουμε την ε, 104 του 2019 μετά από την απόαντηση που θα σταλεί από τη ΣΤΙΟΝ αναφέρονται και στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα ξεκινάμε για το πρώτο σημείο σήμερα το απόγευμα, το σημείο 25 και τώρα θα μιλήσω ισπανικά. Αναφορά 1114 του 2018 από Φιλανδό Επίκο για την ε, υποτιθέμενη ε, βάνευση μεταχείριση των ε, σκύλων στην Κύπρο. Έχουμε εδώ την ανεφέρουσα. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή. Έχετε πέντε λεπτά για να μας εκθέσετε την αναφορά σας και μετά θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μέλη της Επιτροπής και θα έχετε άλλα δύο λεπτά για να κλείσετε την αναφορά σας. Καλωσορίστε, ευχαριστώ και έχετε το λόγο. It's, uh, uh, it's not here. Δεν είναι εδώ. Α, α, εντάξει. Συγγνώμη, συγγνώμη. Νόμιζα ότι είναι εδώ. Ότι έχουμε κάποιους από τους αναφέροντες για αυτή τη συγκεκριμένη αναφορά. Να δώσω λοιπόν απευθείας τον λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Γενική Διεύθυνση Σάντε, Κίρστεν Βόρχαγκεν. Καλημέρα σας. Και ευχαριστούμε πολύ που εδώ ως Επιτροπή έχουμε τη δυνατότητα να εκφράσουμε την άποψή μας και να σας δώσουμε κάποιες βασικές πληροφορίες. Όσον αφορά την αναφορά αυτή, πρόκειται για την ε, υποθέμενες παραβιάσεις προστασίας ε, των ζώων, αδέσποτων σκύλων συγκεκριμένα, στην Κύπρο. Και θα ήθελα να σας πω εδώ ότι το ΕΦΖΙΝ ε, των ε, αδέσποτων ε, ζώων δεν υπόκειται στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εμπίπτει στην αρμοδιότητα των χωρών μελών και μόνον. Η συνθήκη τρόπο εργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα το άρθρο 13 αυτή τη συνθήκη, υποχρεώνει κυρίω τι χώρε μέλη να υπακούν ε, στις απαιτήσει για ο ευζήν την ευμερία των ε, ζώων. Ε, το άρθρο 13 δεν ισχύει για τομείς όπου δεν υπάρχει νομική βάση για την εναρμόνιση σε σχέση με την προστασία των ζώων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγγνώμη, λέει η πρόεδρος, μπορείτε να μιλάτε λίγο ε, βραδύτερα. Να επαναλάβω λίγο μιλήτρια, όχι. Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά την ε, αρμοδιότητα που έχουν αναλάβει βάσει των συνθήκων ε, να μην την υπερβούν, να μην υπερβούν τα όρια αυτής της αρμοδιότητας. Και με το σκεπτικό αυτό η Επιτροπή όσον αφορά την εν λόγω αναφορά δεν, πρόκειται να προβεί στην, δεν θα προβεί στη λήψη μέτρων. Ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν για ε, τα εκώστα ζώα δεν ισχύουν ε, διατάξεις προστασίας των ζώων, αλλά αποκλειστικά διατάξεις περί υγείας στον κτηνιατρικό τομέα. Αυτό σημαίνει δηλαδή διατάξει σε σχέση για, για εμβολιασμό προφύλαξης όσον αφορά την ε, λύσα. Και πάλι για να συνοψίσω, ε, λόγω των περιορισμένων δυνατήτων νομικών ειδικών δυνατοτήτων που έχει στα χέρια της η Επιτροπή, η δημερία, η καλή διαβίωση των ε, ζώων εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των χωρών μελών. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ε, θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Αφού ακούσαμε λοιπόν την Επιτροπή, Λυπάμαι, δεν σας είχα δει. Κυρία Ντανούκα, έχετε το λόγο. Ναι, η, Επιτροπή είπε στην απάντησή της ότι δεν υπάρχει αρμοδιότητα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά την προστασία των αδέσποτων. Αλλά και πάλι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια συνθήκη σε σχέση με αυτό το θέμα, συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και αφορά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Κατοικιδίων, η οποία έχει υπογραφεί από 18 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου υποθέτω ότι υπάρχει δυνατότητα και θα ήταν ευταίο εάν η Επιτροπή στην ε, φάση της ε, εξέτασης της αυτών των αναφορών, γιατί δεν είναι μόνο μια τέτοια αναφορά, αλλά είναι περισσότερες αναφορές που προέρχονται από πολλές χώρες. Ε, παρακαλείται λοιπόν η Επιτροπή να εξετάσει το πώς το εργαλείο αυτό ε, δουλεύει στο επίπεδο του Συμβουλίου της Ευρώπης και τι είδους αξιολόγηση έχει γίνει ούτε ώστε να έχουμε κάποιες πληροφορίες για τους μηχανισμούς παρακολούθησης και για το πώς ε, η σύμβαση αυτή ε, υλοποιείται από ορισμένες χώρες μέλη ούτως ώστε να έχουμε μια διασυνοριακή έποψη του προβλήματος και να το θέσουμε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα ναι, της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω να μην ε, κλείσει η αναφορά αυτή, αλλά να ζητήσουμε από την Επιτροπή την ε, διεξαγωγή μιας περαιτέρω έρευνας και ενδεχομένως την επαφή με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τους αρμόδιους αξιωματούχους που είναι υπεύθυνοι για την ε, εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Ωραία λοιπόν. Καθώς δεν υπάρχει άλλη παρέμβαση, εάν συμφωνείτε, θα μείνει ανοιχτή η αναφορά και θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να μας ενημερώσει για τα θέματα αυτά. Να σας κάνω μια ερώτηση. Σε σχέση με αυτή την αναφορά, λέει η Πρόεδρος. Μάλιστα. Είστε αναφέρουσα. Όχι. Τότε θα πρέπει να συνεχίσουμε. Είστε αναφέρουσα μιας άλλης αναφοράς. Ωραία, θα πάρετε το λόγο. Λοιπόν, η αναφορά αυτή παραμένει ανοιχτή, ούτω ώστε η Επιτροπή να μας ενημερώσει σε σχέση με τα θέματα αυτά της ε, ευημερίας των ζώων. Και τώρα θα περάσουμε στην αναφορά 1868 κάθετος 2014 του Wolfgang Arnold από τη Γερμανία σε σχέση με τη θανάτωση των αδέσποτων στην ε, Ρουμανία και την αναφορά 1484 κάθετος 2016 από τον Μυρκέα Σερμπανόιου της, από τη Ρουμανία εν σχέση με την κακομεταχείριση, ε, κακομεταχείριση συγγνώμη, αδέσποτων στη Ρουμανία. Η Μαρία Βασί ε, η οποία είναι δικηγόρος ε, θα πάρει το λόγο για να υποστηρίξει αυτές τις αναφορές. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε το, την Επιτροπή και μετά θα κλείσει πάλι η κυρία Βασί. Ευχαριστώ πολύ θα σας ε, μιλήσω, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να σας πω ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε εδώ, καταρχάς, και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που μας δώσετε τη δυνατότητα να βρεθούμε εδώ σήμερα. Να σας πω ότι ως εκπρόσωπος ε, της ε, Ομοσπονδίας μας, επειδή ε, στο άρθρο 2 της Συνθήκης εγγυόμαστε τις ε, αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε και την προστασία αξιοπρεπούς ε, ζωής για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική αυτή που εφαρμόζεται για τα δέσποτα είναι μια πολιτική η οποία είναι ενταγμένη στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι Βρισκόμαστε στο 2020, είμαστε ελεύθερα άτομα, είμαστε αξιοπρεπή άτομα, έχουμε όμορφες ζωές και δεν θα μπορούσαμε να παραγνωρίσουμε ότι υποφέρουν ζώα γύρω μας. Πώς μπορούμε να μιλάμε για τη δική μας ευημερία ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ε, βλέπουμε να υποφέρουν σκυλιά ε, λόγω κακομεταχείρισης ε, στη Ρουμανία. Δεν θέλω να προσβάλλω φυσικά την γίνει λογική σας, αλλά θα ήθελα λίγο να δείτε πόσο βάναυση είναι η συμπεριφορά στα ζώα στη Ρουμανία δεν υπάρχουν ε, λύσεις ε, για τα δέσποτα σκυλιά στη Ρουμανία και γιατί αυτό, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, όπως άκουγα και στο παρελθόν και πραγματικά δεν πίστευα ότι θα άκουγα κάτι τέτοιο και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να εξετάσει κατά πόσον ευημερούν ή όχι τα ζώα. Όχι, είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι όταν υπογράφει κανείς τη συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας λέγεται και ότι θα έχουμε φυσική και συναισθηματική ασφάλεια και θα μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι δίπλα στην οικογένειά μας. Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο όταν βλέπουμε γύρω μας ε, και διαπιστώνουμε τέτοιες βάναυσες ε, πράξεις ε, κατά των σκυλιών. Θα ήθελα κάποιον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μας πει ότι σήμερα πρέπει να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να νομοθετήσουμε. Έχετε δικαίωμα να νομοθετήσετε. Δεν έχει μεγάλη σημασία αν είναι υγιή τα ζώα ή ασθενή. Βάσει της ε, προστασίας ε, μιας ε, ψευδονομιμότητας, μιας επίφασης νομιμότητας, επιχειρήσεις παίρνουν πάρα πολλά χρήματα για να θανατώνουν αυτά τα ζώα. η ε, νοοτροπία τους είναι να συλλαμβάνουν και να σφάζουν αυτά τα ζώα. Πραγματικά δεν υπάρχει κοινοτικό δίκαιο, δεν υπάρχει κάτι που να προστατεύει τα ζώα αυτά και στη χώρα μου δεν υπάρχουν αποτελεσματικά μέτρα που να επιτρέψουν σε δικηγόρους να καταγγείλουν αυτές τις ε, αδικίες, αυτές τις βιαιότητες και φρικαλαιότητες. Και πραγματικά ε, θα ήθελα να σας ζητήσω να ευχαριστείτε το Θεό, διότι είστε ευτυχισμένοι άνθρωποι. Αλλά πρέπει πραγματικά να φροντίσουμε και αυτά τα ευαίσθητα ε, όντα, τα ζώα αυτά. Πρέπει πραγματικά να... Ε, δώσουμε συγχαρητήρια στην ε, Πορτογαλία και στη Γαλλία που κατηγοριοποίησαν τα ζώα ως τρίτη κατηγορία ατόμων. Θα ήθελα να συγχαρώ τις χώρες αυτές ε, που έχουν απαγορεύσει τη σφαγή των ζώων. Ε, την Ελλάδα, την Τσεχία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και άλλες χώρες. Είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματικά θέλουμε να ζούμε με την ίδια συναισθηματική ασφάλεια που προσφέρεται και απολαμβάνουν οι πολίτες αυτών των χωρών. Οι Ρουμάνοι θα ήθελαν και αυτοί να είναι περήφανοι που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς λόγω αυτού. Στη Ρουμανία πριν από τρεις εβδομάδες η Κριστίνα Τοπέσκου, μια δημοσιογράφος, πέθανε. Γιατί, διότι όπως και πολλοί από εμά ενεπλάκει στη φροντίδα δεκάδων τέτοιων ζώων για να μπορέσει να αντισταθμίσει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν νομοθετικά και κοινωνικά μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Η γυναίκα αυτή πραγματικά ε, δεν μπορούσε να αντέξει ε, το γεγονός ότι υπέφεραν αυτά τα ζώα. Εσείς είστε εδώ για να νομοθετήσετε. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να σας παρουσιάσω όλο το υλικό που έχω φέρει θα σας τα παρουσιάσω αν θέλετε. Έχουμε πάρα πολλές ε, ταινίες που θα μπορούσατε να δείτε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που μου διαθέσατε. Σκεφτείτε λίγο τις αρμοδιότητές σας. Μπορεί να υπάρχουν αρμοδιότητες και στο γραπτό υλικό υπάρχουν και ε, βάσιμοι λόγοι οι οποίοι στηρίζονται και νομικά ώστε η Επιτροπή Αναφορών να προσπαθήσει να κάνει κάτι και να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να ε, νομοθετήσουν επί του ζητήματος. Δεν είμαστε απομονωμένοι από αυτά τα ζώα τα οποία χρειάζονται προστασία διότι θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία για την ευημερία των ζώων αυτών, η οποία συνάδει και με την ευημερία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Η Κίρστεν ε, Βορχάγεν έχει και πάλι το λόγο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση της, ε, των αναφορών. Κατ' ουσία δεν μπορώ παρά να επαναλάβω τα όσα είπα προηγουμένως, που βεβαίως η Επιτροπή γνωρίζει ότι η κατάσταση προστασία των αδέσποτων ζώων στην Ρουμανία είναι ενδεχομένω προβληματική και μετά από τις περιγραφές που ακούσαμε ασφαλώς και είναι βάση των περιγραφών που ακούσαμε εδώ. Αλλά για να επαναλάβω τα όσα είπα προηγουμένως, η ευημερία των αδέσποτων ζώων δεν ρυθμίζεται από διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει την απαραίτητη νομική βάση προκειμένου να πάρει τα σχετικά μέτρα. Αυτό εμπίπτει στην κάστο αρμοδιότητα των, της χώρας μέλους. Όσον αφορά το άρθρο 13, το οποίο επεσήμενα προηγουμένως, που αφορά τον τρόπο εργασίας για την, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει τις διατάξεις και τις νομικές ε, βάσεις για την ανάληψη δράσης στον τομέα της προστασίας των ζώων. Το άρθρο αυτό λέει τα εξής κατά, την, ε, ε, κατά τον, ε, τη διατύπωση και εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της γεωργίας, της αλίας, των μεταφορών, της εσωτερικής αγοράς, της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της έρευνας στο διάστημα αναλαμβάνουν η Ένωση και οι χώρες μέλη την ευθύνη για τα ζώα ως ε, ε, αισθανόμενα όντα. Και οι χώρες ε, μέλη ακολουθούν βεβαίως θρησκευτικά ήθη, παραδιώσεις και την κληρονομιά τους ε, στοιχεία που αποτελούν την ε, κληρονομιά για την νομοθετική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά δεν περιλαμβάνουν την ε, δράση σε σχέση με την προστασία δάσποτων ζώων. Και στο βαθμό αυτό η Επιτροπή αυτή δρά σύμφωνα με τη νομική βάση και τις συνθήκες που έχουν υπογράψει συμβαλόμενες χώρες μέλη. Ε, άλλα θέματα που δεν εμπίπτουν εδώ εναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των χωρών μελών. Και επιτρέψατε μου να αναφέρω τη σύσταση ε, του Συμβουλίου. Η Επιτρόπη δεν έχει υπογράψει τη σύσταση αυτή, ούτε είναι μέλος. Μέλη είναι χώρες μέλη. Άρα η Επιτροπή και στο πλαίσιο αυτό δεν έχει τις νομικές δυνατότητες να παρέμβει. Η Επιτροπή, η Επιτροπή ωστόσο ε, είναι ενεργή στον τομέα αυτό. Υποστηρίζει για παράδειγμα ε, τον ε, οργανισμό για τη διεθνή καταπολέμηση των ε, ζωονόσων και ο οργανισμός αυτός ε, σε σχέση με την ε, ανάγκη μιας κατάλληλης και παρκούς διαχείρισης των αδέσποτων έχει διατυπώσει κάποια κριτήρια για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου των αδέσποτων ζώων ε, και ε, τα κριτήρια αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τη διατύπωση της σχετικής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο για, την, για τον έλεγχο των αδέσποτων και την άμβλυνση των προβλημάτων που προκαλούν τα δέσποτα σκυλιά στην, ε, στις χώρες μέλη. Η κάθε χώρα θα πρέπει ως πλήρες μέλος ε, του οργανισμού αυτού, ωστόσο, θα πρέπει να λάβει μόνη της την απόφαση πώς θα εφαρμόσει τις ε, διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές στο εθνικό πλαίσιο. Η Επιτροπή υποστηρίζει το έργο του οργανισμού αυτού και τις ε, εργασίες των χωρών μελών, αλλά, επαναλαμβάνω και πάλι, δεν έχει την νομική αρμοδιότητα να ε, θεσπίσει εφαρμοστέο δίκαιο. Συνοπτικά, η ευημερία των αδέσποτων δεν εμπίπτει στο ε, τομέα του άρθρου 13 της Συνθήκης, άρα λοιπόν δεν ε, υπόκειται στις διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή δεν είναι νομικά αρμόδια να παρέμβει στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Κύριε Στοργάρη έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια πράγματα. Ξέρω τις παραμέτρους που έθεσε στην προηγούμενη αναφορά η Επιτροπή και τώρα και για την επόμενη κιόλας, διότι πάλι για ρουμανική περίπτωση αναφορά με θέματα αδέσποτα είναι η επόμενη. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Η συμπεριφορά έναντι των αδέσποτων και των ζώων συνολικότερα είναι ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα με το θέμα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Το θέμα στη Ρουμανία έχει δύο παραμέτρους. Ένα, τις αρχές και τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές ε, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό και το άλλο είναι η ευθύνη των πολιτών και ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι από αυτούς τουλάχιστον αντιμετωπίζουν το ζήτημα. Έχουμε περιπτώσεις όπου υπάρχουν εγκαταλελειμμένα, παρατημένα ζώα στο δρόμο και καταλήγουν εν τέλει σε καταφύγια ή θανατώνονται. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι υποστηρίζω την ιδέα να μείνει η αναφορά αυτή ε, ανοιχτή και να υπογραμμίσουμε εκ νέου τις καθηγητές γραμμές του Συμβουλίου. Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Ζντάνοκα να αντιμετωπίσουμε, να απευθυνθούμε στο Συμβούλιο για να ζητήσουμε ε, περαιτέρω εμπλοκή ε, του Συμβουλίου και πληροφορίες και από τις Ρωμανικές Αρχές. Δεν νομίζω ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος με ομότητα, με βαναυσότητα είναι ε, ευρωπαϊκή συμπεριφορά και αυτό αφορά και τις Ρουμανικές Αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, είναι αδιανόητη μια τέτοια βαρβαρική συμπεριφορά, ιδίω όταν ασκείται σε ένα κράτος μέλος της Ένωσης. Στην Βουλγαρία, τη χώρα μου, οι, σφαγή και, οι σφαγές και οι ακροτηριασμοί ζώων τιμωρούνται με φυλάκιση. Η Κομισιόν λέει ότι το άρθρο 3.13 ε, δεν της δίνει αρμοδιότητες. Έχει αρμοδιότητες όμως σε άλλους τομείς. Την καταχώρηση των ζώων συνοδείας. Αν δεν υπάρχει μηχανισμός ε, ευρωπαϊκός θα υπήρχε μικρότερο, μεγαλύτερος έλεγχος, ε, μικρότερος έλεγχος των αδέσποτων και μικρότερη προστασία των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεχίζουμε να μην έχουμε το, το νομοθετικό πλαίσιο για το εμπόριο των ζώων συνοδείας και αυτό σημαίνει ότι τα ζώα αυτά μπορεί οποτεδήποτε να ε, βρεθούν στο δρόμο. Πρέπει να υπάρξει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο ούτω ώστε τα ζώα να αντιμετωπίζονται με ανθρώπινο τρόπο. Αλλιώς δεν θα κάνουν τίποτα ούτε οι υπόλοιποι. Πιστεύω λοιπόν ότι η, αναφορά πρέπει να μείνει ανοιχτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σντάνοκ έχει το λόγο. να πω δύο λόγια για αυτά που είπε η Επιτροπή στη δεύτερη αναφορά της. Λέτε ότι δεν υπάρχει νομοθετική δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Εμείς όμως από την Επιτροπή θέλουμε όχι μόνο διαβουλεύσεις, αλλά και πιο ενεργή δράση. Είστε εδώ οι διαμεσολαβητές μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης και των νομοθετών. Αν το Συμβούλιο της Ευρώπης μπορεί να δεχθεί μια σύμβαση για την προστασία των ζώων συνοδείας, γιατί δεν μπορεί να το κάνει ένα αντίστοιχο η Ευρωπαϊκή Ένωση. με νέα νομοθετικά κείμενα. Αυτό προτείνω. Είναι μια ευρωπαϊκή σύμβαση εύλογη, 18 κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών Κύπρος, Λιθουανία, η Ρουμανία. Έχουμε πολλές δυνατότητες να εξετάσουμε πώς λειτουργεί το εργαλείο αυτό και να μάθουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη δική μας ε, νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο Νούμπο μπορεί να γίνει, ε, θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων των Ανθρώπων. Γιατί να μην δει και άλλες συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης όπως αυτό για την προστασία των ζώων συνοδείας. Ναι, αξιόλογη κυρία Προ... αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, θα ήθελα να αναφερθώ ε, στις ε, αναφορές ε, αυτές που αφορούν τα ζώα. Ε, επιτέλους έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Ε, όλες τις αναφορές έχουν συγκεντρώσει πάνω από 80.000 υπογραφές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, στράτευση υπέρ των ζώων. Ανεξάρτητα από το αν ε, πρόκειται για ε, σκυλιά τα οποία ε, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο κυνήγι αλλά τελικά κακοποιούνται βάναυσα ή αδέσποτα τα οποία θανατώνονται βάναυσα στη Ρουμανία. Ε, δεν είναι δυνατόν ε, ενώπιον των φερμένων αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση να μείνει άπραγη. Και στη Βουλγαρία η αντιμετώπιση των αδέσποτων είναι απαράδεκτη. Μετά τον ευνοχισμό ε, τα ζώα αυτά αφήνονται ελεύθερα στο δρόμο, στη μοίρα τους ή μένουν σε κάποια κέντρα κλεισμένα μέχρι το τέλος της ζωής τους ε, ανάπηρα ε, ζώα ή απλώς περιτά ζώα θανατώνονται. Ε, άρα λοιπόν στο τομέα αυτό θα πρέπει να υπάρξουν εναρμονισμένοι κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δάσποτα παλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους. Τα χτυπούν αυτοκίνητα, τα σκοτώνουν, πεθαίνουν από την πείνα ή πεθαίνουν από διάφορες ασθένειες. Σε ορισμένες χώρες ε, μοιάζει να είναι εθνικό σπορ να κυνηγάνε αυτά τα ταλέπορα ζώα. Η λύση δεν μπορεί να ισοδυναμεί με θανάτωση. Οι ενδιαφερόμενες ε, χώρες, οι οποίες πλήττονται από ένα μεγάλο αριθμό δέσποτων ζώων, ε, θα πρέπει να έχουν ε, προγράμματα εμβολιασμού και στήρωσης. Σήμερα ψηφίστηκε ένα σημαντικό ε, ψήφισμα για το εμπόριο, παράνομο εμπόριο ζών. Ε, το ψήφισμα αυτό θα επιτρέψει και μια καλύτερη αναγνώριση των ε, αδέσποτων και σήμανση των αδέσποτων ζών. Θα παρακολούσα λοιπόν οι αναφορές αυτές που αφορούν τα αδέσποτα ζώα να παραμείνουν ανοιχτές. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά στην αναφέρουσα για να κλείσει. Ευχαριστώ όλους σας που γιατί καταλαβαίνετε το θέμα που θέτω. Να σας θυμίσω τα εξής. Το ψήφισμα 2016 του 12 που περιέχει σύσταση προς το, του Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή για να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των ζώων. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 12. Τίποτα πέραν της σύστασης. Κανείς δεν σε εμποδίζει να αναλάβετε να λάβετε μέτρα. Σας παρακαλώ λοιπόν πραγματικά με κάθε σεβασμό να μην μας ξεχάσετε. Ο πόνος των ζώων αυτών συνεχίζεται. Το ότι δεν τον βλέπετε στις Βρυξέλλες δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Εξ ονόματος λοιπόν των ζώων αυτών σας ζητώ νομοθετήστε, έχετε την αρμοδιότητα. Δείτε όλο το γραπτό υλικό μας. Δεν μπορούσα να μιλήσω για όλο το γραπτό υλικό. Εκεί όμως υπάρχουν λύσεις που προτείνονται αστυνομία ζώων ως επίσημη υπηρεσία, μια επίσημη υπηρεσία της Ρουμανίας. Δείτε τα κείμενά μας για να, για να γίνουν πραγματικοί Ευρωπαίοι πολίτες ή Ρουμάνοι πρέπει να λυθούν τα προβλήματα αυτά. Αν δεν γίνει κάτι γι' αυτό, ε, δεν θα γίνουν πραγματικοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάστε αντικειμενικά την κατάσταση στην Ρουμανία. Μας βοηθήσατε να γίνουμε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βοηθήστε μας να αλλάξουμε τα πράγματα στη χώρα. Γιατί ο πόνος είναι τεράστιος μεταξύ των ζώων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ακούσαμε την αναφέρουσα, την Επιτροπή, τα μέλη της Επιτροπής μας. Προτείνουμε να μείνει ανοιχτή η αναφορά και ζητούμε θα στείλουμε μια επιστολή στο Συμβούλιο στο Συμβούλιο της Ευρώπης ζητώντας Τέλο πάντων, θα ενημερώσουμε το Συμβούλιο τη Ευρώπη για τι αναφορέ που υπάρχουν για την ε, κακή συμπεριφορά κατά των ζωών, ε, την έλλειψη ε, αρμοδιότητας και νομοθετικής ρύθμισης στο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα τονίζοντας ότι είναι δική τους ευθύνη να αναφέρουν στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει τη σύμβαση αυτή πολλά από τα οποία είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιμένουμε λοιπόν από το Συμβούλιο να μας απαντήσει για την αναφορά αυτή. Ευχαριστούμε. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Σημείο 27. Αναφορά 475 του 2016 της Γκαμπριέλα Παπαντόποβα, βουλγαρικής ηθαγένειας, εξ ονόματος μιας σειράς εταιριών προστασίας ζώων, ζώων με άλλες 464 υπογραφές για την ε, αδιαφορία έναντι των ε, αδέσποτων σκύλων στη Βουλγαρία. Θα δώσω πέντε λεπτά στην ε, κυρία Γεωργίευα που μίλα εξ ονόματος αναφέρουσας και στο τέλος έχει και δύο λεπτά για να κλείσει. Ευχαριστούμε και καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα, να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω την αναφορά αυτή εξ ονόματος 18 ενώσεων προστασία ζώων στη Βουλγαρία, από όλη τη χώρα. Η αναφορά μας ανατρέχει στο 2016 αφορά την αντιμετώπιση των αδέσποτων σκυλιών και των ε, ζώων ε, συνοδείας στη Βουλγαρία και την έλλειψη αποτελεσματικής νομοθεσίας από πλευράς κράτους για να λύσει το πρόβλημα. Αρχικά, οι προσφυγίες μας συνοδεύονταν από αυτές τις εικόνες που έδειχνε τις άθλιες συνθήκες των χώρων ε, των καταφυγίων για τα ζώα, τα οποία μόνο καταφύγια δεν είναι, γιατί εκεί τα ζώα πεθαίνουν από ασυτεία, από κρύο, από ασθένειες. Η εθνική δομή που είναι υπεύθυνη για την προστασία και την εφαρμογή της νομοθεσίας προστασίας των ζώων, η Υπηρεσία Ασφάλειας των Τροφίμων της Βουλγαρίας δηλαδή δεν ασκεί πραγματικό έλεγχο. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το ότι οι αρχές της Βουλγαρίας όχι μόνο αντιβαίνουν στην εθνική νομοθεσία, αλλά παραβιάζουν συστηματικά και το άρθρο 13 της, Ευρωπα... της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπηρεσία αυτή στη Βουλγαρία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή ενός τεράστιου σώματος νομοθετικών κειμένων και στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας. Η αδυναμία της έχει επιπτώσεις και πέραν των εθνικών συνόρων. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες, διότι το 2018 όταν συζητήθηκε εδώ η αναφορά μας, λάβαμε μεγάλη υποστήριξη από την πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή Αναφορών. Δυστυχώς λόγω τεχνικών λόγων δεν υπήρχε αρκετός, χρόνο, χρόνος, δεν έγινε επίσκεψη κατανόησης της κατάστασης. Το πρόβλημα τώρα όχι μόνο συνεχίζει να υπάρχει, επιδεινώθηκε και όχι μόνο στη Βουλγαρία. Απόδειξη είναι ότι αντίστοιχη με τη δική μας ε, αναφορά έχουν κατατεθεί από Βουλγαρία, Ιταλία, από Ιταλία, Ισπανία κλπ. Στην Βουλγαρία τα αγαθά, που, τα, τα ζώα που αγοράζονται και πολλούνται δεν ελέγχονται. Δεν υπάρχει υποχρέωση ούτε καταγραφής αλλά ούτε καν ε, εμβολιασμού. Στα σπίτια, στα περισσότερα σπίτια, σπίτια στην Βουλγαρία ε, τα σκυλιά ε, ε, συνοδεύουν τα αυτοκίνητα όπως βλέπετε. Αν κάνετε μία έρευνα Google στη Βουλγαρία θα δείτε πάνω από 5.000 αποτελέσματα πώληση, για πώληση των, των ζώων. Ένα, ένα μόνο site όχι μόνο περιλαμβάνει πωλήσει ζώων αλλά και αγώνες μεταξύ σκύλων που είναι αδίκημα. Σε μία έρευνα της Deutsche Welle πέρσι ε, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ε, παράνομη πώληση εκατομμυρίων σκύλων σε όλη την Ευρώπη από διάφορες τοσεβίδε τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία κυρίως. Αυτό το εισόδημα το, ε, για, από την εμπορία ζωών είναι αντίστοιχο με το ύψος του εισοδήματος από ναρκωτικά γύρω στα 24 δις ευρώ το χρόνο. Οι ερευνητέ λένε ότι τα περισσότερα ζώα είναι σε πολύ άθλια κατάσταση και πεθαίνουν πολύ γρήγορα. Γι' αυτό ανησυχούμε ιδιαίτερα για την παράμετρο υγιεινής και ασφάλεια και δημόσιας υγείας. Όχι μόνο για τις χώρες από όπου προέρχονται τα ζώα, αλλά και για τις χώρες στις οποίες πηγαίνουν. Οι πολιτικές αυτές δεν σέβονται άλλωστε το διατάξεις του άρθρου 13. Μια άλλη έρευνα του BBC πέρσι δείχνει ότι η Βουλγαρία έχει γίνει κέντρο δικτύου αγώνων σκύλων σκυλό, ε, ε, από όλο τον κόσμο. Οι ερευνητέ είπαν ότι, ρητά, ότι βρήκαν ένα παράνομο εμπόριο από την Ανατολική Ευρώπη μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία. Ταυτόχρονα η Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων της Βουλγαρίας έστειλε μια επιστολή δύο χρόνια πριν την έρευνα στην ίδια επιτροπή το ίδιο, για την ίδια αναφορά που, εξε, που και είπε ότι όλη η παράνομη πρακτική αγώνων σκύλων έχει σταματήσει. Θυμίζω ξανά ότι η υπηρεσία αυτή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή ενός τεράστιου όγκου ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Μετά από χιλιάδες μηνύματα προς όλες τις ε, ε, αρμόδιες αρχές, μαζικές διαδηλώσεις και αποφάσεις δικαστηρίων δεν έχουμε καν σε εθνικό επίπεδο υλοποιήσει αυτές την, αυτή την νομοθεσία με αποτέλεσμα πανευρωπαϊκά ε, πανευρωπαϊκές συνέπειες. Ζητούμε λοιπόν εκ νέου από εσά να επανεξετάσετε το ενδεχόμενο να επισκεφθείτε την Βουλγαρία και να συνεχίσετε να ασκείτε πίεση προς τις βουλγαρικές αρχές. Η Επιτροπή είχε κομβικό ρόλο στην υιοθέτηση του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου για την εφαρμογή και υλοποίηση και υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για το θέμα. Έτσι εκφράζεται πραγματικά αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες της Ένωσης. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η αναφορά μας είναι επίκαιρη και μπορεί να λάβει νομοθετική πλαισίωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την κυρία Φορχάγεν. Um, ευχαριστώ πολύ. Και σας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δέσμευσή σας και ε, ας ξεκινήσουμε με την ε, παράκληση που διατυπώσετε στο τέλος. Όσο ε, μένουν ως έχουν οι συνθήκες, η Κομισιόν δεν έχει δυναμική βάση ε, να προβεί σε νομοθετικό ψήφισμα. Αυτό το οποίο κάνει όμως η Κομισιόν είναι εκούσια μέτρα και τα εφαρμόζει πράγματι ε, σας ε, μίλησα προηγουμένως για τον ε, αρμόδιο οργανισμό. Υπάρχει μια πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ζώων, η οποία συστάθηκε το 2017 από την Κομισιόν και η οποία προσφέρει τη δυνατότητα μιας ε, ανταλλαγής και βασίζεται σε κούσιες πρωτοβουλίες των ενδιαφερόμενων. Και εδώ υπάρχει επίσης και μια εκούσια πρωτοβουλία για την προστασία σκύλων και γάτων. Η ψηφιακή αυτή πλατφόρμα αυτή τη στιγμή διατυπώνει, επεξεργάζεται μάλλον συστάσεις και προηγουμένως αναφερθήκατε στην ε, διαδικτυακή εμπορία και για το θέμα αυτό επεξεργάζεται κάποιες συστάσεις για πολιτές μέσω του ίντερνετ αλλά και για ε, operators των, από τις διάφορες πλατ, ε, των, ε, στις διάφορες πλατφόρμες του ίντερνετ ε, προκειμένου να τους την προσοχή σε ζώα τα οποία πολλούνται μέσω ίντερνετ, κατά πόσο είναι νόμιμο το εμπόριο, κατά πόσο έχουν εμβολιαστεί, κατά πόσο έχουν το, την ελάχιστη επιθρεπτή ηλικία κλπ. κλπ. Η εφαρμογή όλων αυτών των πραγμάτων, για να το επαναλάβω, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των χωρών μελών εδώ η Επιτροπή δεν μπορεί παρά να προσφέρει τη δική της συνδρομή και δυνατότητες στήριξης. Ε, τον Αύγουστο 2018 ε, ψήφισε μια σύσταση κομισιών βάσει της οποίας ε, θα πρέπει οι χώρες μέλη να ελέγξουν τις πλατφόρμες στο διαδίκτυο προκειμένου να δουν πώς διαμορφώνεται η κατάσταση με την ε, πώληση ε, σκύλων και γάτων ή την προσφορά. Ε, τέλος του 18, αρχές του 19, συμμετείχαν 17 χώρες αυτή την αξιολόγηση, συν Ελβετίας παρατηρήτρια και αποκαλύφθηκαν ε, κάποια προβλήματα και ορισμένοι πάροχοι ε, σε ορισμένες πάροχους επιβλήθηκαν ε, κάποιες κυρώσεις. Λήφθησαν κάποια μέτρα σχέση με αυτούς. η νομική βάση για την σύσταση αυτή εκ μέρους της Επιτροπής είναι... αφορά τις εκούσιες αυτές πρωτοβουλίες. Δεν, δε δεν υπάρχει νομική βάση ή κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, για Κομισιόν έχει επίγνωση του προβλήματος και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της να υποστηρίξει τις χώρες μέλη. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. I'm going to speak in Maltese. Um... Ο κύριος Σαλίμπα, θα μιλήσω μαλτέζικα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι δυνατόν να έρχεται να μας λέει ότι δεν έχει αρμοδιότητα για τα καταφύγια για τα ζώα. Ναι, μεν το καταλαβαίνουμε, αλλά όπως ακούσαμε και από την αναφέρουσα και θα ήθελα να την ευχαριστήσω προσωπικά για την επιμονή της μας είπε για τη διακίνηση ζώων από τη Βουλγαρία και από άλλα κράτη-μέλη. Στην ενιαία αγορά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι μπορεί να κάνει συστάσεις και μόνο και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Όταν έχουμε ζώα τα οποία μεταφέρονται από τη μία χώρα στην άλλη και πολλούνται από τη μία χώρα στην άλλη. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ θεωρώ απαράδεκτο. Ε, θεωρώ ότι πλέον έχει φτάσει η κατάλληλη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νομοθετήσει για τη μεταφορά ζώων τα οποία πολλούνται, ακόμα και αν αυτό γίνεται μέσω διαδικτύου. Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα και να μην ε, απλώς εκδίδουμε συστάσεις, διότι οι συστάσεις πρέπει να εφαρμόζονται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι εφαρμόζονται. Επομένως, ε, θα ήθελα να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και ελπίζω να έχουμε πολύ πιο συγκεκριμένη δράση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν γίνεται πώληση ζώων από τη μία χώρα μέλος ε, στην άλλη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σντάνοκα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπα και προηγουμένως για το ενδεχόμενο να κάνουμε κάτι χρησιμοποιώντας και τους μηχανισμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Υπάρχει και μηχανισμός παρακολούθησης και εποπτείας. Για αυτή τη συγκεκριμένη αναφορά θα ήθελα να ευχαριστήσω την αναφέρουσα και όλους τους ανθρώπους, τους 464 που υπέγραψαν την αναφορά και για την επιμονή τους και για την επαναλαμβανόμενη ε, αναφορά στην Επιτροπή μας και το γεγονός ότι προτείνεται να γίνει ε, αποστολή στη Βουλγαρία. Λυπάμαι, δεν θα μπορέσουμε να πάμε ε, ε, για να δούμε επιτόπου τι γίνεται με τη συγκεκριμένη αναφορά, αλλά μπορούμε να βρούμε ίσως λίγο χρόνο να μιλήσουμε μαζί σας στη Σόφια, όπου θα γίνει η αποστολή. Ελπίζω να υπάρξει λοιπόν περαιτέρω συνεργασία και εξακολουθώ να πιστεύω ότι η Επιτροπή θα είναι πιο δραστήρια στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ράντεφ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ είμαι βέβαιος ότι αυτή η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή Στην ε, Βουλγαρία έχουμε σίγουρα προβλήματα ακόμα με τα ζώα συντροφιά ε, και με τα δέσποτα σκυλιά που εγκαταλείπουν ο κόσμο στο δρόμο και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα δέσποτα σκυλιά και γάτες που έχουμε στο δρόμο. Τα τελευταία χρόνια η Βουλγαρία έκανε πολλές προσπάθειες ε, για να επιλύσει το πρόβλημα. Στι τελευταίες ε, τροπολογίες τη νομοθεσία για την προστασία των ζώων, για παράδειγμα το 2010, εισήχθηκε η έννοια του Εθνικού προγράμματο ε, για μια σειρά από μέτρα για να μειώσουν τον αριθμό των σκύλων που είναι αδέσποτα και ε, σε κάποιους δήμους ε, γίνεται δουλειά, σε κάποιες άλλες δεν γίνεται τίποτα. Το θέμα είναι ότι ε, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για τα μέτρα αυτά. Πρέπει καταρχάς να ευαισθητοποιούν οι κάτοχοι ζών συντροφιά, ώστε να είναι πιο υπεύθυνοι και να αναλαμβάνουν πραγματικά τα ζώα τους. Ε, και επίσης να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τον οριθμό των ζώων που είναι εγκαταλελειμμένα. Δυστυχώς ε, εγκαταλείπονται πολλά ζώα ε, και από την άλλη ζώα τα οποία βρίσκονται στο δρόμο πρέπει να λαμβάνουν και αντιπαρασιτοκτόνο αγωγή και να μπορούμε να τους επιστρέφουμε και στις περιοχές καταγωγής τους για να μην έχουμε ε, και ε, εισβολή νέων ζώων. Για παράδειγμα, όταν μειώνεται ο αριθμός των ε, σκύλων και αρουραίων, αυξάνεται ο αριθμός των γάτων. Επομένως, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να αντιμετωπίσουμε το πρόγραμμα. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ γενικό. Στο μέλλον θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα από τους διάφορους δήμους και βασίζομαι και στην καλή βούληση του κάθε Δήμου και ελπίζω να βρουν κοινού τρόπου μαζί με τι φιλοθροπικέ οργανώσει που βρίσκονται σε κάθε Δήμο. Είναι πάρα πολύ δραστήριε οργανώσει αυτέ, οι φιλοζωικέ, συγγνώμη, και πρέπει να μπορέσουμε να. Στη Βουλγαρία έχουμε περίπου 25 ε, εγκαταλελειμμένους ε, Στη Σόφια, για παράδειγμα, έχει μειωθεί τρεις φορές ο αριθμός των ζώων από 11.400 το 2007 Φτάσαμε στις 3.000 ζώα. Υποτριπλασιάστηκε λοιπόν ο αριθμός ε, μέσα σε 10 χρόνια. Θα πρέπει να ευχαριστήσω και πάλι τους αναφέροντες ε, για το γεγονός ότι έφεραν ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα και το γεγονός ότι είναι τόσο δραστήριοι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των εγκαταλελειμμένων ζώων. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, ώστε οι αρμόδιες αρχές στη Βουλγαρία και ο οργανισμός ε, και όλοι οι κατάλληλοι φορείς να κάνουν όλες τις προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον ε, αριθμό των ε, καταλελειμμένων ζώων και να βρούμε μία λύση στα προβλήματα των ε, καταλελειμμένων ζώων για τα ζώα συντροφιάς. Θα πρέπει να συνεχίσουν να κάνουμε ελέγχους και να επιμείνουμε ώστε όλα τα νόμιμα μέτρα να γίνονται σεβαστά όσον αφορά την ευημερία των ζώων. Εγώ προσωπικά δεσμεύομαι ώστε να επιμείνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ομάδα Εργασίας Προστασίας των Ζώων, στην οποία είμαι αντιπρόεδρος, ώστε τα θέματα αυτά να αναλύονται καταλήλως και να προσπαθήσουμε τελικά να ε, έχουμε και ένα νόμιμο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία των ζώων συντροφιάς και των εγκαταλειμμένων ε, ζώων, των αδέσποτων. Ε, τέλεια. Η αναφέρουσα τώρα έχει δύο λεπτά. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. El señor... Συγγνώμη, ο κύριος Κρίστοφ. Ε, κυρία Πρόεδρε, οι εικόνε που, που είδαμε και τα όσα μα είπατε είναι πραγματικά ιδιαίτερος βάναυσε. Το 2018 ε, εγκρίναμε ένα ψήφισμα το οποίο ε, κάνει έκκληση προς την αστυνομία προκειμένου να εκπονήσει μια στρατηγική για τα δέσποτα ζώα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση του Συμβουλίου Ευρώπης. Παρ' αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να, πάρουμε, να λάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες ή ε, να εγκρίνουμε μια σχετική νομοθεσία. Επίσης, η πρόταση θέσπισης νομοθετικού πλαισίου είναι μια καλή πρόταση. Τα προβλήματα των αδέσποτων, ιδιαίτερα στη Βουλγαρία, συνιστούν πρόβλημα που σχετίζεται με την ε, διαφθορά και πιστεύω ότι θα ήταν καλό να επισκεφθεί τη Βουλγαρία μια αποστολή προκειμένου να εξετάσει το πρόβλημα αυτό από πολλές, ε, βάσει πολλών ε, οπτικών προσεγγίσεων. Και η αναφορά θα πρότεινα να παραμείνει ανοιχτή. Ο κύριος Λαβάκοφ. Ευχαριστώ. Να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο. Δυστυχώς η αναφορά αυτή διατυπώθηκε και ετοιμάστηκε με, πιο, με πολύ γενικό τρόπο και πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένη. Η αναφορά περιλαμβάνει κάποια πράγματα με τα οποία δεν συμφωνώ. Δεν υπάρχει ρεκόρ εκτροφή σκύλων αγώνων. Παντού υπάρχουν προβλήματα με ε, τα σκυλιά και ιδίω τα δέσποτα σκυλιά. Δεν είναι μόνο θέμα της Βουλγαρίας και της ε, Ρουμανίας. Στις Βρυξέλλες δεν υπάρχει τίποτα ζωντανό ζώο. Αυτό με έχει εντυπωσιάσει από τότε που ήρθα. Ούτε, ούτε κουνούπια δεν βρίσκεις. Στην ε, Ρώμη μπορεί να δείτε χιλιάδες εγκατατελειμμένες ε, γάτες. Ε, δεν υπάρχει πρόβλημα με τα ζώα αυτά. Είναι συνηθισμένα, συνηθισμένος ο κόσμος. Το πρόβλημα είμαστε εμείς, δεν είναι τα ζώα. Πρέπει να... Προφανώς δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση όπως τώρα. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιες περιοχές ε, της Σόφιας για παράδειγμα υπάρχει ένα πρόβλημα με τα αδέσποτα. Άνθρωποι είμαστε, κάποιος πρέπει να τα φροντίσει, πρέπει να, τα, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά τους, αλλά αυτό απαιτεί μια ευρύτερη νομοθετική ρύθμιση. Ευχαριστώ. Η αναφέρουσα έχει δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής που έδειξαν κατανόηση στα θέματα που θέτουμε. Προτείνω εκ νέου να επισκεφθείτε την Βουλγαρία. Ακόμα περισσότερο είναι αναγκαίο, διότι ο κύριος ε, ο έχει κάποιες επιφυλάξεις για την ε, κατάσταση. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω την ανυπόφορη αντιμετώπιση κατάσταση των ζώων, ιδίω των ε, ζώων συνοδείας, που οδηγεί σε δυσαρέσκεια των πολιτών έναντι των οποίων είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε την αναφέρουσα. Την ευχαριστούμε που ήρθε μαζί μας. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής. Προτείνουμε να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Και πράττουμε ό,τι και για την προηγούμενη. Θα στείλουμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης τις αναφορές αυτές για την ευημερία των ζώων, ιδίως για τα σκυλιά τα δέσποτα σκυλιά, ζητώντας από το Συμβούλιο να ασκήσουν πίεση στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τη σύμβαση που έχουν υπογράψει. Επόμενο σημείο. 82-2018 αναφορά από ένα άτομο λιθουανικής ηθαγένειας για την αδιαφορία των δημοτικών αρχών του Κλαϊπέντα σε θέματα και σε περιπτώσεις ε, βάναυση συμπεριφοράς ε, έναντι ζώων. Είναι εδώ οι αναφέρουσες. Ποιος από τους δυο θα μιλήσει. Ποια από τις δυο θα μιλήσει. Και οι δύο, μία, δύο άτομα. Συνολικά έχετε πέντε λεπτά. Και στο τέλος συνολικά δύο λεπτά. Μπορείτε να το μοιραστείτε όπως θέλετε. Πέντε λεπτά συνολικά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, κάθε χρόνο οι δήμοι στη Λιθουανία σκοτώνουν δεκάδες χιλιάδες ζώα με δημόσιους διαγωνισμούς, με εμπορικέ ε, επιχειρήσεις, νουάρους, μεντράγια και άλλους. Αυτές οι συμφωνίες ε, χρηματοδοτούνται από δημόσια κονδύλια που μεταξύ των ε, Λιθουανών αποκαλούνται στρατόπεδα συγκέντρωσης των ζώων. Είδατε τις φωτογραφίες των ζώων στην αναφορά μας. Παρά την, ε, τις διαμαρτυρίες των πολιτών, οι πρακτικές συνεχίζουν για πάνω από 20 χρόνια. Τα κράτη-μέλη έχουν τοπική ευθύνη για την, ε, έχουν τοπική νομοθεσία για την ε, προστασία των ζωών, αλλά από ό,τι φαίνεται είτε είναι πολύ ανεκτικοί οι νόμοι, είτε παραβιάζονται συνεχώς. Δεν συμφωνούμε με την Κομισιόν ή το άρθρο 13 τη Συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ο κύριος Αντρουκάητης, πρώην Επίτροπος, είχε υπογραμμίσει τότε στην κυρία Βίξτρομ ότι στην παλιότερη αναφορά μας ότι πολιτική του προτεραιότητα, πολιτική μου προτεραιότητα το Σαντοκαρής ως υπεύθυνο επίτροπο για την ασφάλεια και την, των τροφίμων και για τη θέματα υγείας, η ασφάλεια. Καταλαβαίνω τη σημασία της ευημερία των ζώων για τους πολίτες της Ένωσης. Επίσης γνωρίζουμε ότι η ευημερία των ζώων είναι ένα μόνιμο θέμα στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών και απαιτεί και δείχνει μόνιμη ανησυχία των πολιτών και αναφερόντων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του στις 4 Ιουλίου του 2012 για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων από το 2012 στο 2015 είχε καταγράψει ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ευημερία των οικόσιτων ζώων. Το Κοινοβούλιο υπογράμμιζε την ανάγκη, την επίκουσα ανάγκη να υπάρξει ένα πλαίσιο, ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ευημερία των ζώων και πρότεινε λεπτομεριακές συστάσεις για την εφαρμογή συγκεκριμένων προτάσεων ε, για ένα νόμο πλαίσιο συνένωση. Εσείς είπατε το ανάποδο. Τι από τα δύο ισχύει. Ιδού η απορία που πρέπει να απαντηθεί. Uh, <clears throat> uh, we also ask the Commission The new Η νέα επιτροπή που ξεκίνησε να λειτουργεί πρέπει να αναλύσει βαθύτερα την αρμοδιότητα της Ένωσης για το άρθρο 13. Πολλά προβλήματα, πολλές αναφορές υπάρχουν για το θέμα αυτό. Άρα υπάρχει ανάγκη δράσης της Ένωσης. Ζητούμε να μην κλείσετε την αναφορά, να λάβετε μέτρα για να υιοθετηθεί ένα νομικό πλαίσιο για τα ζώα συνοδείας. Μέχρι τότε οι Ευρωπαίοι είναι ίδιοι με τους άγριους που τρώνε αυτά τα ζώα. Ζητήθηκε δράση από το Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση της παράνομης αγοραπολισίας ζώων, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, θέλουμε κι άλλο συνεχίζει. Υπάρχει μεγάλη ομότητα έναντι των ζώων στο επίπεδο της νομοθεσίας. Αυτή η συμπεριφορά επικυρώνεται από συμφωνίες μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και δήμων, παραβιάζοντας το άρθρο 13 της Ειδικής Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ συχνά η νομιμότητα απέχει πολύ από την ηθική στη χώρα μας. Δεν μπορεί να είναι επιλεκτική η νομιμότητα και επιλεκτική η ηθική πρέπει να υιοθετηθεί ένα νομικό πλαίσιο που θα δείχνει ότι πηγαίνουμε προς μία επίλυση του προβλήματος. Ε, αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ένωσης, Γερμανία, Ρουμανία, Κύπρος και αλλού. Όλοι στην ίδια κατάσταση βρισκόμαστε. Κρατήστε ανοιχτή την αναφορά και προσπαθήστε στο βαθμό που γίνεται να συμπεριλάβετε τον ίδιο πληθυσμό και σε συμβάσεις που δεν έχουν ήδη προστατευτεί από την Ένωση ή υιοθετήστε νέες συμβάσεις για τα αδέσποτα. Γάτες, σκυλιά που τα πετάνε οι ιδιοκτήτες τους στο δρόμο και που πρέπει να προστατευθούν. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά ζητάμε να αναλάβετε δράση. Ζητάμε να ασκήσετε πίεση, να οργανώσετε κάποιες μελέτες και να μην κλείσετε την αναφορά. Muchísimas gracias. Ahora tendría la palabra la comisión, la señora Kirsten. Και τώρα ο λόγο στην Επιτροπή, στην κυρία Φορχάκη. Ευχαριστώ πολύ. Από τα όσα είπαν οι αναφέροντες, σχημάτισα την εντύπωση ότι ίσως έχει δημιουργηθεί μια παρανόηση το άρθρο 13 το άρθρο 13 της συνθήκης είναι η νομική βάση για την θέσπιση διατάξεων, νομικών διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για διατάξεις προστασίας των ζώων, αλλά μόνο για τους ε, τομείς που αναφέρονται εκεί και οι τομεί αυτή δεν περιλαμβάνουν την προστασία των αδέσποτων ζώων. Το άρθρο 13 βεβαίως δίδει τη δυνατότητα ε, θέσπισης νομικών διατάξεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για άλλους τομείς, όχι για τα αδέσποτα ζώα, για άλλους πολιτικούς τομείς. Ε, Κύλοι και γάτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χρήση τους για εμπορικούς στόχους ε, εμπίπτουν στις ε, σχετικές διατάξεις του εμπορίου, της εμπορίας ε, ζώων. Υπάρχει σχετική οδηγία υγείας που αφορά το θέμα αυτό. Αυτή η νομική βάση αφορά ε, ζητήματα όπως είναι ο προληπτικός εμβολιασμό κατά της λύσης η ε, διατάξη γυνής όσον αφορά την ε, διατήρηση των ζώων ή την μεταφορά τους. Όσον αφορά τα δέσποτα, επαναλαμβάνω και πάλι, λέει ο Μιλήτρια, δεν μπορούμε να εκδώσουμε νομικές διατάξεις από την Κομισιόν ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ να κάνω μία διόρθωση. ήθελα μόνο να επισημάνω το εξή. Η νομική διάταξη στην οποία ήθελα να αναφέρω δεν είναι οδηγία αλλά κανονισμός. Αυτός ε, σημαίνει ότι ισχύει ε, ε, για όλες τις χώρες μέλη και είναι η παριθμόν 576 του 2013 και αφορά τη διατήρηση κόστων ζώων για σκοπούς άλλους από αυτούς της, ε, του εμπορίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος ε, από την Επιτροπή το λόγο. Κανείς. Ωραία. Να δώσουμε το λόγο για δύο λεπτά στις αναφέρουσες. Εμείς ζητούμε, ζητούμε ειδικά για τα αδέσποτα ζώα, να συμπεριληφθούν στο άρθρο 13 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι είναι ε, ζώα και επομένως είναι όντα και θα πρέπει να αναφέρεται ο όρος αδέσποτα ζώα, stray animals. Επίσης, περιμένουμε και ζητούμε την υποστήριξή σας και εκτιμήσαμε και ιδιαίτερο τη βοήθειά σας και εκτιμούμε και την υποστήριξη και των άλλων κρατών μελών και των υπολείπων αναφερομένων που βρίσκονται εδώ σήμερα και θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει, μάλλον από την Επιτροπή σας, να έρθουν στη Λιθουανία για διερευνητική αποστολή γιατί πραγματικά θα εκπλαγείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, στις αναφέρουσες για τη σημερινή τους παρουσία εδώ. Μετά από τα όσα ακούσαμε και από τα όσα ακούσαμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μιας και συζητήσαμε και αρκετές αναφορές σήμερα το απόγευμα για την ε, κακομεταχείριση των ζώων, η πρόταση της Προεδρίας είναι να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και σε αυτό το πακέτο προτάσεων ε, για όλες τις αναφορές για τα δέσποτα και εγκαταλελειμμένα ζώα και την κακομεταχείριση των ζώων θα θέλαμε να αποτανθούμε στο Συμβούλιο και επομένως τα αφήνουμε ανοιχτό μέχρι να λάβουμε απάντηση. Για την τελευταία αναφορά, γιατί πάντα θέλω να εξηγώ ε, για το τελευταίο σας αίτημα ε, στους αναφέροντας να γίνει αποστολή της Επιτροπής Αναφορών και να έρθουμε να δούμε τι γίνεται στη Λιθουανία. Ε, οι συντονιστές είναι οι αρμόδιοι, οι εκπρόσωποι της κάθε κοινοβουλευτικής ομάδος και από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα αποφασίσαμε για όλες τις αποστολές του 2020. Είναι ήδη λοιπόν καθορισμένες οι αποστολές που θα γίνουν φέτος και Επομένως θα πρέπει ε, να γίνει το αίτημα σε οποιαδήποτε πολιτική ομάδα για το 2021 για να γίνει μια τέτοια αποστολή. Ε, δεν είναι μοναδική αρμοδιότητα της Προεδρίας να αποφασίζει για το αν θα γίνει μια αποστολή ή όχι. Ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρουσία και αποφασίζουμε φυσικά να παραμείνει ανοιχτή η αποστολή. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Σημείο 29, αναφορά 823 του 2013 από τον κύριο Σάχερ γερμανικής ε, ηθαγένειας για τις νομικές διατάξεις που επιτρέπουν τη θανάτωση ζώων στη Δανία. Νομίζω ότι δεν είναι εδώ αναφέρον, επομένως να δώσω το λόγο στην Κομισιόν, στο Γενική Διεύθυνση Σάντε και στην κυρία Χίρστεν Φον Χάγκεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Äh, äh, και εδώ δεν μπορώ παρά να επισημάνω και πάλι αυτά τα οποία ήδη έχω πει. Και εδώ η Επιτροπή δεν έχει την ε, δυνατότητα να αναλάβει δράση. Και εδώ θα ήθελα να σας παραπέμψω στις κατευθυντήριες ε, γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων η οποία έχει εκδώσει, ο οποίος έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του πληθυσμού των αδέσποντων σκύλων και επίσης να σας επισημάνω ότι η καταχώρηση των αδέσποτων και ο έλεγχος γεννήσεων των αδέσποτων είναι η βάση μιας υπεύθυνης ε, διαχείρισης ε, αυτών των πληθυσμών. Ε, βεβαίως ε, παράλληλες προσεγγίσεις για τον έλεγχο των ε, αδέσποτων πληθυσμών των σκύλων ε, θα πρέπει να εφαρμοστούν και η θανάτωση των αδέσποτων σκύλων δεν θεωρείται βιώσιμη στρατηγική. Ε, στις προδιαγραφές θα πρέπει να περιληφθούν ε, ανθρώπινες ε, μέθοδοι για τη διαχείριση αυτών των πληθυσμών. Παρ' όλα αυτά, εναπόκειται στις χώρες μέλη, ως πλήρη μέλη αυτού του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων, να ελέγξουν το πώς θα εφαρμόσουν τις, κατευθυντήριες, τις ε, παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές βάσει των εθνικών τους δεδομένων και προϋποθέσεων. Η Κομισιόν πρόκειται να θα συνεχίσει να συνδράμει το έργο αυτού του οργανισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος ε, το λόγο από τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών. Όχι. Παρακαλώ. Ähm, Ευχαριστώ πολύ. Μόνο στην συντομία θα ήθελα να πω το εξή και εγώ θα ήθελα να συστήσω όπως και με διαδικασία που ακολουθήθηκε στις άλλες αναφορές και, για, και ως προς την αναφορά αυτή να μείνει ανοιχτή παρακαλώ. Ναι, ευχαριστούμε πολύ και εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι η Δανία είναι μεταξύ των 18 χωρών μελών που είναι μέλη της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και ίσως θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω διερευνήσεις του θέματος. Πρόταση είναι λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να ζητηθεί από την Επιτροπή να δοθούν γραπτές απαντήσεις εφόσον η αναφορά αυτή δεν έχει αποσταλεί προς την Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά θα θέλαμε να επιληφθούμε. Να επιληφθείτε και να μας διαβάσετε μια γραπτή απάντηση. Ε, Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης αφορά την αναφορά 443 κάθε 2018 του Μάρκο Τζιοβανέλη από την Ιταλία που περιλαμβάνει 80.000 ε, υπογραφές εκ μέρους του Future 4 Wildlife ε, σε σχέση με την έγκριση ειδικής νομοθεσίας για την προστασία και τη διαχείριση των ζώων συνοδείας, κατοικιδίων και αδέσποτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, στην αναφορά 0167 2017 από τον κάτοικο της Κύπρου KJ ε, για την ε, σύσταση μιας ε, υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να είναι επιφορτισμένη με την ευημερία των ζώων και αυτό χωρίς καθυστέρηση. Παρακαλώ, ε, εκπροσωπείτε την αναφορά υπαριθμών 0167. Έχετε πέντε λεπτά να μας παρουσιάσετε το θέμα, κυρία Φάλκον. Α, όχι. Λέγομαι ε, Κάθριν... Α, Γεωργαλή. Ε, και κάθε φορά που επισκέπτομαι την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο και την Ιταλία, διαπιστώνω ότι υπάρχουν χιλιάδες αβοήθητα ζώα. Μπορώ να συναισθαθώ την, ε, τον πόνο τους και ε, αισθάνομαι ακόμα μεγαλύτερη οδύνη σήμερα ακούγοντας ότι δεν υπάρχει καμία νομική βάση για την προστασία αυτών των ζώων. Αυτό με θλίβει βαθύτατα και θα ήθελα να προτείνω στον Οργανισμό για την Ευημερία των Ζώων να βοηθήσουν τα ζώα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως είπε ο Μαχάτμα Μαγκάντι, το μεγαλείο ενός έθνους μπορεί να ε, αποδειχθεί από τον... να φανεί στον τρόπο που μεταχειρίζεται τα ζώα. Εμείς ε, έχουμε αποτύχει παταγωδός, δεν έχουμε φανίσει απολύτως καμία τέτοιου είδους μεγαλειώδη ε, αντιμετώπιση των ζώων τα ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται θύματα βάναυσης ε, μεταχείρισης. Είδαμε τις ε, φωτογραφίες αυτές. διασμένες γάτες. Βλέπουμε πολλές τέτοιες στην Ελλάδα και στην Κύπρο. ακόμα και άγρια ζώα. Πώς μπορεί κανείς να αφαιρθεί σε ένα άγριο ζώο με αυτόν τον τρόπο. Αυτό δείχνει κάτι για τον χαρακτήρα αυτών των ανθρώπων. Και μου λέτε ότι δεν υπάρχει νομαθεσία προκειμένου να προστατευτούν τα ζώα αυτά. Αυτό ήταν εξαιρετικά θλιβερό. Πώς μας ε, επηρεάζει. Ε, τέτοια άρρωστα ζώα βρίσκονται παντού, ε, στους φούρνους, στα σπίτια μας κλπ. Πλήττεται και ο τουρισμός. Ε, κάθε φορά που έρχονται τουρίστες ε, ε, κάθε φορά που πάω διακοπές σε ένα νησί, εάν δεν ξαναβρω τις γάτες που γνώριζα, είναι γιατί έχουν φάει φόλα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βασίζεται σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άτομα, ιδιώτες, οι οποίοι καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά στο Facebook και ζητούν πόρους. Τι κάνουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, απολύτως τίποτα. Στην καλύτερη περίπτωση ε, φυλακίζουν ε, τα ζώα και μετά τα αφήνουν ελεύθερα και δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν κάποιοι πόροι για αυτές τις ΜΚΟ ε, που έχουν πολύ συχνά ποσά, γελιότητες δηλαδή, 3.000 ευρώ το χρόνο. Το RSPCA είναι ο παλαιότερος οργανισμός ε, για τα ζώα. Συστάθηκε πριν από 200 χρόνια στο, στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρόκληση ε, να αναγνωρίσει το κοινό ότι τα ζώα δεν είναι ε, άψυχα όντα, αλλά πλάσματα με συνέστηση. Ε, για παράδειγμα, πώς μεταχειρίζονται τους ε, γαϊδάρους, τους χρησιμοποιούν για... Ε, τους εκμεταλλεύονται και όταν δεν είναι πλέον σε θέση να επιταλέψουν την εργασία τους, τους σκοτώνουν, τους πετάνε από τον κρεμό σε κάποιες χώρες. Και δεν υπάρχει καμία νομική βάση για την προστασία αυτών των ζώων. Ο Οργανισμός για την Ευημερία των Ζώων στην Ευρώπη προτείνει να δημιουργηθούν ε, παρόμοιες υποδομές προς την RCPCA, να ε, δημιουργηθούν τέτοια κέντρα ε, σε κάθε χώρα, κατάλληλοι χώροι, στελεχωμένοι με προσωπικό, προκειμένου να διασώζονται τα ζώα από τους δρόμους και να τους παρέχουν προστασία. Επίσης, υποστήριξη παρέχεται και στο πλαίσιο του Εράσμους, όπου μπορούν ε, οι φοιτητές της κτηνιατρικής ε, να βοηθήσουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους οι ΜΚΟ και εθελοντές ε, όπως εγώ η ίδια. αυτό δεν στοιχίζει πολύ τίποτα στους Ευρωπαίους πολίτες, κάτι σαν 10 δολάρια το χρόνο και επίσης ο οργανισμός αυτός της ευημερίας των ζώων στην Ευρώπη μπορεί να επισκεφθεί σχολεία και να κάνει ενημερωτικές εκστρατείες για τους μαθητές προκειμένου να κατανοήσουν ότι τα ζώα είναι... θα πρέπει να προστατεύονται. Θα ήθελα να σας αναφερθώ ένα εδώ σενάριο όπου παιδιά μεγαλώνουν σε χώρους όπου εξοικειώνονται ακόμα και με γουρούνια, με αλεπούδες κλπ. Τα άτομα είναι ζώντα πλάσματα, δεν είναι αντικείμενα, χρειάζονται τροφή, χρειάζονται περίθαλψη, στοργή κλπ. Θα σε ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Κομισιόν. Η κυρία Κέστεν Φόχαγγιν, παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. και πάλι. Επιτρέψατε μου να σας πω κάτι το οποίο εσείς ίδια μόλις είπατε. Ε, ποτέ δεν είπα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει νομοθεσία για την προστασία των ζώων. Υπάρχει μία νομοθεσία για την προστασία των ζώων τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των χωρών μελών. Αυτό το οποίο εγώ είπα είναι ότι για, τον τομέα, για, τα αδέσποτα ζώα εδώ δεν υπάρχει νομική βάση για την Ευρωπαϊκή, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να παρέμβει. Για τα αδέσποτα αυτή η αναφορά ε, δεν θα πρέπει να αναφέρεται μόνο στα δέσποτα. Γι' αυτό θα ήθελα να παραπέμψω στρατηγική για την προστασία των ζώων, η οποία έχει ψηφιστεί το 2012 έως το 2015 όπου είχαν προβλεφθεί ποικίλα μέτρα προκειμένου να εφαρμοστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα ήθελα να σας επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τη στρατηγική αυτή προκειμένου να διευκρινίσουμε ε, τι είδους επιπτώσεις είχε η στρατηγική αυτή και σε ποιο βαθμό έχει εφαρμοστεί. Και υποθέτουμε ότι τα αποτελέσματα θα τα έχουμε μέχρι το τέλος του χρόνου και στη βάση αυτών των αποτελεσμάτων θα δούμε τι είδου περαιτέρω μέτρα θα πρέπει ενδεχομένως να προταθούν ή να ληφθούν. Εμείς από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορούμε να αλλάξουμε το άρθρο 13 των συνθήκων. Εμείς ε, μπορούμε να βασιστούμε, να βασίσουμε τις εργασίες μόνο στην, ε, στις νομικές βάσεις των συνθήκων, όπως είπα ήδη κατ' επανάληψη. Ε, τι, α, κατά πώς υπάρχουν κάποιες άλλες δυνατότητες, εδώ δεν μπορώ να πω κάτι. Άρα λοιπόν, θα περιμένουμε, θα αναμένουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και βεβαίως στο πλαίσιο της νέας ε, Επιτροπής του Νέου Σώματος θα ε, διατυπωθούν οι νέοι στόχοι του έργου της Επιτροπής. Αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι προβλέψιμα τα αποτελέσματα. Αλλά όπως σας είπα, στον ορίζοντα αυτό ε, τοποθετώ την αναφορά αυτή του σημείου 30. Ευχαριστώ. Ο λόγος στα μέλη τώρα. Ο κύριος Σαλίμπα. Ναι, δεν σχολίασα κάθε αναφορά, διότι νομίζω ότι οι περισσότερες είναι αντίστοιχες. Όμως το πρόβλημα αυτό της προστασίας των ζώων είναι σαφές, είναι σαφέστατα τα όσα βλέπουμε εδώ στην Επιτροπή μας την τελευταία ώρα. Πρόκειται για ένα συστηματικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει σε μια σειρά από κράτη-μέλη. Στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Κύπρο. Πρόκειται λοιπόν για υπαρκτό πρόβλημα, απτό πρόβλημα. Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες αφιερώνουν ώρες από το χρόνο τους σε εθελοντική εργασία, επενδύουν τα ίδια τους τα χρήματα για να μπορέσουν να βελτιώσουν κάπως την κατάσταση και κάθε φορά που ακούω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφέρεται σε αρμοδιότητες, περιορισμούς ε, και όρια, ε, εξανίσταμε. Πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι πολύ πιο δημιουργική, να πιέσει τα κράτη-μέλη. Συζητούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό τι πρέπει να γίνει, αλλά στην πραγματικότητα οι πραγματικέ λύσει για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, για να υπερασπιστούμε αυτά τα ζώα που δεν έχουν φωνή, χρειάζονται εμά για να τα προστατεύσουμε, δεν υπάρχουν. Ε, δεν έχουμε ακούσει κάποια λύση. Επιμένω λοιπόν, η αναφορά αυτή πρέπει να παραμείνει ανοιχτή ιδανικά εμείς ως Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να κάνουμε αποστολές σε όλες τις χώρες που αναφέρθηκαν, διότι είναι κρίμα να βλέπουμε τέτοιες φωτογραφίες, αλλά πρέπει πλέον να περάσουμε και από τη θεωρία στην πράξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τα μέσα και πρέπει να ε, χρησιμοποιήσει περισσότερο τη δημιουργικότητά της, ε, διότι έτσι θα μπορέσει να πιέσει και τα κράτη-μέλη. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη φρικτή κατάσταση ε, που βιώνουν αυτά τα ζώα. Ευχαριστώ τον κύριο Σαλίμπα. Η κυρία Εύη έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να παρέμβω και εγώ για αυτές τις αναφορές για να εκφράσω εν γέννη την υποστήριξή μου ε, στα όσα ακούσαμε σήμερα το απόγευμα και ιδιαίτερα στις τελευταίες αναφορές, διότι το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο έχει αρχίσει να λαμβάνει σίγουρα σημαντικές διαστάσεις. Ε, αναφέρονται πάνω από 100 εκατομμύρια ζώα, αδέσποτα ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τα οποία είναι εκτεθειμένοι σε κακομεταχείριση και σε κάθε ε, μορφής ε, βίαιης συμφοράς και πολλές φορές ε, τα συλλαμβάνουν και τα χρησιμοποιούνται ως πειραματόζωα σε εργαστήρια, χρησιμοποιούνται στα καλλιντικά ή και είναι και κρέατα για σφαγή, τα οποία χρησιμοποιείται κατά την εκπαίδευση των σκύλων που χρησιμοποιούνται σε μάχες και ορισμένες φορές είναι και στην κατάσταση και εξολοθρεύονται ολόκληροι πληθυσμοί αδέσποτων ζώων. Πρόκειται για κάτι το οποίο πρέπει κάπως να το αντιμετωπίσουμε και κατά την άποψή μου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι σε κάποιες χώρες αυτό το θέμα έχει γίνει πλέον ε, κατεπήγον και υπάρχουν και συνέπειες και για την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων και για κάποια είδη ε, τα οποία είναι προστατευόμενα είδη και αυτοί οι δύο τομείς είναι τομείς αρμοδιότητας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μέχρι τώρα όμως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας επαναλαμβάνει συνεχώς ότι δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία και ότι δεν υπάρχει τρόπος να παρέμβουμε αλλά είναι εκατοντάδες οι αναφορέ ε, που ακούμε εδώ στην Επιτροπή των Αναφερών για το θέμα αυτό. Υπάρχουν χιλιάδε πολίτε οι οποίοι ζήτησαν να δοθεί κάποια λύση, κάποιο τέλο ε, σε αυτή τη μάστιγα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα το οποίο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, κάνει μια νομοθετική πρόταση για να υπάρχει ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν προσπαθεί να παρακολουθεί κινήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει. Και υπάρχει και μία ε, πρόταση της Επιτροπής Αναφορών ε, η οποία ε, καταγράφει ότι το θέμα είναι επίγον και πρέπει να γίνει κάτι. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρύβεται πίσω από ένα φύλλο σικής, το φύλλο της εθνικής αρμοδιότητας. Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν περιθώρια δράσης και αν υπήρχε η πολιτική βούληση να δράσει κάποιο, θα μπορούσαμε να κάνουμε τεράστια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ελπίζω πραγματικά ότι η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δείξει τελείω διαφορετικό προσανατολισμό σε σχέση με την προηγούμενη και να αποφασίσει επιτέλου να τίνει ευήκονου ε, στα όσα λένε οι χιλιάδε πολίτε για να σταματήσει αυτή η μάστογα στο θέμα αυτό. Και θα ήθελα κι εγώ, όπω και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, να ζητήσω να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και να σταλεί μαζί με τα πρακτικά ε, της σημερινή συζήτηση στη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επανεξέταση. Ελπίζω επίσης ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Green Deal όπου το θέμα τη της ευημερίας των ζώων επιτέλου εύχομαι ότι θα λάβει περισσότερο χώρο, θα υπάρχει και η δυνατότητα να δράσουμε από αυτό και το οφείλουμε πάρα πολύ ε, σίγουρα στους πολίτες και στα ζώα τα οποία ε, αξίζουν να μην υποφέρουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Εύη. Και τώρα έχετε δύο λεπτά για να ολοκληρώσετε για την αναφορά 167. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φον Χάγεν είπε ότι υπάρχουν νόμοι, αλλά όχι για τα δέσποτα ζώα. Εγώ αναφέρομαι στα δέσποτα ζώα. Άρα δεν υπάρχει τίποτα για να τα προστατεύσουμε αυτά τα ζώα. Ποιος μπορεί να κάνει κάτι για να δημιουργήσει αυτού του νόμου. Εγώ δεν μπορώ, δεν είναι δική μου δουλειά. Κάποιο πρέπει όμω ε, να νομοθετήσει. Εγώ δεν έχω έρθει εδώ για πλάκα. Έχω έρθει γιατί ελπίζω ότι θα μπορέσω να τα βοηθήσω γιατί δεν έχουν φωνή. Ποιο έχει φωνή, ποιο είναι αυτό ο οποίο μπορεί να νομοθετήσει. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια κατεύθυνση γιατί εγώ χρειάζομαι την καθοδήγησή σας. Τον ελεύθερο χρόνο μου τον προσφέρω. Έχουν ψυχή αυτά τα ζώα εγώ έχω υιοθετήσει 8 ζώα και σταμάτησα να ταξιδεύω στην Ελλάδα και στην Κύπρο για να μην βρω άλλο. Ελπίζω να μπορέσετε να κάνετε κάτι από αυτού. Ζητώ τη βοήθειά σας ε, ταπεινά και είμαι εδώ και θα κάνω ό,τι μου πείτε για να μπορέσουμε να τους δώσουμε φωνή. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Yes. Ευχαριστώ. να τονίσουμε το αίτημα της Επιτροπής για μια νέα αξιολόγηση δεδομένης της νέας σύνθεσης της Επιτροπής και των άλλων δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων το, την Πράσινη Συμφωνία, τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, όπου θα παρέχω θα ε, παρουσιάζονται τα αιτήματα διαφόρων φορέων για τις μελλοντικέ αρμοδιότητες και κοιό, μεταξύ άλλων. Προτείνουμε λοιπόν την Επιτροπή για να προχωρήσει σε περαιτέρω αξιολόγηση. 443. Είναι στην μερίσια διάταξη, δεν υπάρχει αναφέρον. Υπάρχει μια επιστολή του Επίτροπου Αντουκάητης από τις 16 Ιουνίου του 2019 συνεχίζει να λέει ότι δεν υπάρχουν αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τα κρατάμε λοιπόν όλα ανοιχτά και την 443 και να ζητήσουμε από την Επιτροπή αξιολόγηση. Ναι, ωραία. Επόμενο θέμα, το 31 Εξήτα ένα διοθόνη η, η ομιλήτρια του 2019 της Ιζαμπέλα Καβαλέτη Ιταλής για την απαγόρευση της αλίευσης καρχαριών και των προϊόντων που προέρχονται από καρχαρίες. So we have... Ah, petitioner is not here. He's following the web streaming. Δεν είναι παρούσα η αναφέρουσα, παρακολουθεί τη συνάντηση με web streaming. Η Επιτροπή. Η κυρία Ελίζα Ρόλερ. Όχι, Κατραζίνα Τζάνιακ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Εξ ονόματος της Επιτροπής θέλω να σας ενημερώσω για την δράση της Ένωσης για την διαχείριση του είδους των, καθαριών, των ειδών καθαριών μετά από αίτημα της εν λόγω αναφέρουσας. Η αναφέρουσα ανησυχεί λόγω του τεράστιου ρυθμού καρχαριών που αλλιεύονται κάθε χρόνο και οδηγεί σε μεγάλη μείωση του πληθυσμού. Και τονίζει ότι η Ένωση παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην αγορά κρέατος Καρχαρία. Ζητά επίσης μεγάλη διαφάνεια στην παροχή πληροφοριών για την φύση των ε, ψαριών που παρέχονται στην κατανάλωση. Ξεκινώ λέγοντας ότι όλοι γνωρίζουμε πως οι καρχαρίες παίζουν ζωτικό ρόλο για τη διατήρηση της των οικοσυστημάτων της θάλασσας και είναι ευάλωτοι στις ανθρώπινες δραστηριότητε μεταξύ αυτών και της αλίας, όχι μόνο όμως. Επίσης, είναι σημαντική και φθηνή πηγή τροφίμων. Πολλοί κόσμος εξαρτάται από το φαγητό. Υπάρχουν πέντε, πολλά είδη μάλλον ε, ε, καρχαριών που όλα τίθενται σε κίνδυνο. Η μη βιώσιμη πρακτική καθαριώνει, είναι πρόβλημα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί ωστόσο, δεν πρέπει να γνωρούμε ότι είναι πρόβλημα περιορισμένο. Η μεγάλη πλειοψηφία των ε, αποθεμάτων καρχαριών είναι σε καλή κατάσταση. Τι κάνει η Ένωση. Εμείς δεσμευόμαστε υπέρ της βιώσιμης διαχείρισης των ε, καρχαριών όπως και των άλλων βιολογικών έμβριων ειδών. Στην κοινή αλληλευτική πολιτική, η προσπάθειά μας είναι να, ε, να ανακτηθούν να ανακτηθεί ο ρυθμός των αλλιευμάτων και μια, με, με υγιή είδη. Εμείς έχουμε βασικές μια σειρά ε, δράσεων. Πρώτον, προστασία των ε, ε ειδών. Άρα γενική απαγόρευση αλίευση των συγκεκριμένων ειδών. Πολλά είδη καρχαριών προστατεύονται, είτε με όρια αλίευσης είτε με απαγόρευση αλίευσης. Υιοθετήσαμε μία πολιτική για να απαγορευτεί η χρήση των πτεργίων, που είναι ένας βασικός λόγος αλίευσης. Δεύτερον, βιώσιμη διαχείριση των αλιευμάτων. Η αλίευση θα πρέπει να γίνεται με βιώσιμο τρόπο βάσει επιστημονική συμβουλή, Η Ένωση υιοθέτησε μια σειρά τεχνικών μέτρων για την προστασία των διαφόρων ειδών, π.χ. απαγόρευση χρήσης απλαδιών στη Μεσόγειο ή ε, δικτύων ε, πυθμένα, μείωση, για να τη μείωση της, ε, των παραλιευμάτων νέες μορφές επιλεκτικών, καλύτερων ε, αλλιευτικών εργαλείων. Μείωση, ε, αύξηση της έρευνας που σχετίζεται στην, ε, στις οικολογικές ε, δραστηριότητες. Είναι κρίσιμο να επενδύουμε σε επιστημονικά δεδομένα, συλλογή και έρευνα για τους ε, καρχαρίες. Και εδώ χορηγούνται κονδύλια της Ένωσης. 5 εφαρμογή των αρμόδιων διεθνών και εθνικών κανόνων. Οι προσπάθειες μας εδώ έχουν στόχο τη σωστή ε, εφαρμογή των σχετικών κανόνων. Πιστοποίηση της, ε, σημείο 6, πιστοποίηση των ε, αλλιευμάτων. Έχουμε, έχουμε ευρωπαϊκούς κανόνες για την διάφανη και πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών και για την αλλίευση των καρχαριών. Επίσης, η Επιτροπή υπόβαλε μια πρόταση αναθεώρησης ε, του συστήματος ελέγχου αλληλείας για να ενισχυθούν οι σχετικές διατάξεις προστασίας. Επίσης, έχουμε και εργαλεία εμπορικού χαρακτήρα. Οι σάιτες, για παράδειγμα, που προβλέπει την προστασία των απειλούμενων ειδών από την υπερεκμετάλλευση μέσω περιορισμού στο εμπόριο όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια και σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Επιπλέον, η Επιτροπή προωθεί μέτρα προστασίας της αλληλείας βάσει επιστημονικών ευρημάτων μέσω των περιφερειακών αλληλευτικών οργανώσεων όπου η Ένωση είναι μέλος προωθούμε την FNAP, δηλαδή Strict Fins Naturally Attached Policy. Το 2019 ήταν η επέτειος ε, της δράσης της Ένωσης για την διαχείριση ε, και συντήρηση των ειδών ε, καρχαριών και ζητήθηκε να εξετάσουν την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, ιδίως για την αλίευση καρχαριών στην περιοχή. Αυτό θα καθοδηγήσει και τα επόμενα βήματα της Επιτροπής. Με αυτά υπόψη κλείνω ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να υποστηρίξει μία απαγόρευση γενικά της αλίευσης και πώλησης προϊόντων ε, από καρχαρίες, διότι η υφιστάμενη κατάσταση επιτρέπει την αλίευση των περισσότερων ειδών, προστατεύει τα απειλούμενα είδη και το διεθνές εμπόριο παρακολουθείται. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ρύθμιση επαρκής για την εξασφάλιση της νομιμότητας και βιωσιμότητας. Επίσης η Ένωση πιστεύει ότι η Ένωση ε, περιλαμβάνει επαρκή νομοθεσία για την αλίευση και την ενημέρωση που επιτρέπουν στον καταναλωτή να κάνει μια πλήρη επιλογή. Σας διαβεβαιώνω ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει την αξιολόγηση για την διατήρηση του καθεστώτος διατήρησης των βασικών ειδών καρχαρία και να εφαρμόζει μέτρα διαχείρισης της αλίευσής του στην Ένωση και αλλού. Θα παρακολουθεί το εμπόδιο και την ε, αλίευση ανά, ε, ε, ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο με στόχο τη διατήρηση του πληθυσμού των ειδών καρχαρίων. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ζάνιεκ. Συνάδελφοι, κύριος Ντούσμαν, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, κρίμα που δεν μπόρεσαν να παραστούν οι αναφέροντες. Ε, το, η αλεία των καρχαριών ανθίζει. 50 εκατομμύρια ετησίως ε, χάνουν οι καρχαρίες βάναυσα τη ζωή τους ε, για το κρέας τους, αλλά κυρίως για τα πτερίγια τους, τα οποία αποκόβονται ε, ενώ τα ζώα ζουν ακόμα, ρίχνονται πάλι στη θάλασσα που πεθαίνουν ε, με φρικτό τρόπο. Ε, ε, οι οικολόγοι καταδικάζουν αυτές τις μορφές ε, δρυμύτατα. Επειδή έχουν μακρά αναπαραγωγική περίοδο, τα, δεν μπορούν να ρυθμιστούν γρήγορα τα αποθέματα. Η κατανάλωση των πτεργίων οδηγεί στην μείωση των αποθεμάτων. Ε, η Ινδία και η Κίνα δεν είναι οι μόνοι αγοραστές αυτών των προϊόντων και ορισμένες χώρες Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης υποστηρίζουν αυτό το εμπόριο. Εμείς οι άνθρωποι ε, παίρνουμε από τα ζώα αυτά τα οποία θέλουν να χρησιμοποιήσουμε για δικό μας όφελος, χωρίς ε, να σεβόμαστε καθόλου τα ζώα. Εδώ θα πρέπει να μεριμνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των ειδών αυτών και παρακαλούμε η αναφορά να μείνει ανοιχτή. Ευχαριστούμε. Η κυρία Εύη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ απολύτως με το συνάδελφο Μάρτιν, διότι έφυξε ένα από τα σημεία τα οποία πραγματικά με σόκαρε το γεγονός ότι κόβουμε τα πτερίγια, ε, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται ως ε, τροφή για αυτές τις ε, περιβόητες σούπας καρχαρία, ενώ το ζώο το ξαναπετάμε στη θάλασσα όπου βρίσκει ένα βίαιο αργό και πόδινο θάλατο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Πάνω από 300 εκατομμύρια ήδη σκοτώνονται κάθε χρόνο 11.000 την ώρα για διατροφικούς σκοπούς ε, και για πολλούς άλλους λόγους. Και ε, το ζώο αυτό, το οποίο ε, κινδυνεύει όλο ένα και περισσότερο με εξαφάνιση. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα μας ανέφερε ένα κατάλογο με καλές προτάσεις, ε, πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε στο μέλλον, αλλά εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά για να παρακολουθήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των πρωτοβουλειών που θα εφαρμοστούν στο μέλλον, αλλά και επίσης για να θυμόμαστε και εγώ προσωπικά θα συμφωνούσα επίσης ε, να υπάρχει απαγόρευση αλίας ε, καρχαριοειδών και εμπορίας ε, των προϊόντων ε, καρχαρία. Και επίσης σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνει ανοιχτή αναφορά και κυρίως είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να γίνονται πολύ περισσότεροι έλεγχοι, πολύ πιο αυστηροί, μεγαλύτερη διαφάνεια στην τηλεκοθεσία για τα ηχθη προϊόντα, τα αλλιευτικά προϊόντα και επομένως θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, θα πρέπει να το παραπέμψουμε και στην Επιτροπή Αλίας για γνωμοδότηση και για ε, να το γνωρίζει επίσης και η ομάδα για την ευημερία των ζώων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Εύη. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Μιας και τα δύο μέλη της Επιτροπής Αναφορών που έλαβαν το λόγο πρότειναν ε, να παραμείνει η ανοιχτή αναφορά, είχαμε μια αρχική πρόταση να κλείσει, αλλά μιας και υπάρχει μια πλήρης και αναλυτική απάντηση μένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετά πλήρης, ε, διότι τα μέλη έχουν αντιρρήσεις, επομένως ε, έχετε πολλή δουλειά ακόμα. προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια για το θέμα και να μας δώσετε και περισσότερες πληροφορίες και να μας πείσετε ότι δεν ε, υπάρχει απειλή για τους καρχαρίες. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περαιτέρω δράση. Ωραία, δεν βλέπω κάποια αντίρρηση. Και τώρα... 32. Σημείο 32. Γύρισε εκεί πρόεδρος, επομένως να τα πει πια. Παρακαλώ. Estamos a 32, ¿no? Buenas tardes. Ahora estamos en la petición en el Περνάμε στο σημείο 32 της ημερήσιας διάταξης, αναφορά 354 του 2019, από τον Ζωάν Σιμονέτ Πόνς, Ισπανικής ε, Ιθαγένειας, ε, για από την Οργάνωση Νέων Γεωργών ε, των Βαλαιαρίδων Νήσων για την προστασία των πουλιών στις Βαλιαρίδες Νήσους. Να καλωσορίσουμε τον αναφερόμενο και να του δώσουμε πέντε λεπτά για να μας παρουσιάσει την αναφορά του. Μετά θα ακούσουμε μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και μετά θα, έχετε, ε, θα ακούσουμε μετά τα μέλη της Επιτροπής μας και δύο λεπτά για να απαντήσετε. Σας δίνω το λόγο για πέντε λεπτά και καλώς ορίσατε. Μ' ακούτε, ναι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βαλιαρίδες νήσους ε, δεν είμαστε κατά ε, των ε, θεμάτων προστασίας των ζώων. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη βιοπικιλότητα του πλανήτη. Θα είναι λίγοι όμως οι γεωργοί στην Ευρώπη που θα θέλουν να συμμετέχουν σε τέτοια δίκτυο. Ε, δεν απαγορεύεται η παραδοσιακή γεωργική δραστηριότητα όπως επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν βοηθούν και την ανάπτυξη της γεωργίας στις ε, προστατευόμενες περιοχές. Δεν αυξάνεται το γεωργικό εισόδημα και δεν βελτιώνεται η ζωή των γεωργών η παραδοσιακή μορφή της γεωργίας δεν επιτρέπει τον εξυγχρονισμό, νέες υποδομές, αντικατάστασης καλλιέργειας ε, με ε, είδη πιο προσαρμοσμένα στην, αγωγή, στην αγορά και ε, πιο καθαρά ύδατα. Αυτό φυσικά ε, δεν επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες δυνατότητες. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κατάλληλο γεωργικό εισόδημα σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε και αλλαγή σκητάλης από πλευράς γενεάς και εγκατάλειψη των περιοχών και είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρόβλημα αυτό, κυρίως ε, στη Μαγιόρκα. Δεν υπάρχει κανένα επιπλέον ε, όφελος ε, στις περιοχές αυτές τις οποίες δραστηριοποιούνται οι γεωργοί. Και επομένως θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι ε, το να ανακηρύξουμε μια νέα περιοδοστατευόμενη περιοχή για τα πουλιά, θα πρέπει να θεμελιώνεται καταλήλως και να υπάρχει μια κατάλληλη δήλωση που να το τεκμηριώνει ο οργανισμός μας το 2017 ξεκίνησε μια διαδικασία για την ε, ανακήρυξη νέων περιοχών και είχαμε αρκετές περιοχές οι οποίες ήταν γεωργικές, ε, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα θα μπορούσαμε να τις αναπτύξουμε στη Μαγιόρκα. Μέχρι ε, πρόσφατα είχαμε διάφορες περιοχές, ορεινές, θαλάσσιες, χωρίς δυνατότητες ανάπτυξης λόγω των γεωγραφικών χαρακτηριστικών τους. Και υπήρχαν μόνο ε, κάποια στοιχεία τα οποία έχει υπογράψει κάποιο σύμβουλος περιβάλλοντος ε, και δεν υπήρχαν εγγραφά ή επιστημονικέ μελέτε που αναδείκνυαν την αξία για τα πουλιά τα οποία θα έπρεπε να προστατευτούν σε αυτέ τι περιοχέ. Ε, τα όσα δόθηκαν στην κοινωνία των πολιτών ε, αναφερόταν μόνο σε ε, οδηγού ε, και κάποια πράγματα τα οποία είχαν γίνει το 2001 και το 2003, κάποιες μελέτες και έλεγε για παράδειγμα το 2016 ε, ένα ζευγάρι ε, ανέτρεφε πουλιά κοντά στις ε, πληγήσεις περιοχές και κάποια ορνηθολογικά στοιχεία χωρίς καμία επιστημονική υποστήριξη. Αναφέρονται για παράδειγμα είδη που δεν είναι σε κίνδυνο, όπως οι φραγκόκοτες. Και επίσης αναφέρονται και κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για τα πουλιά, τα οποία καθορίζονται από το «Cyber Life και πρέπει να πω ότι ε, δεν υπάρχουν κάποια είδη τα οποία είναι τόσο σημαντικά όπως λέει η έκθεση που έστειλε η Επιτροπή ε, στην Επιτροπή σας. Ε, ο καθορισμός κάποιων ε, περιοχών είναι παράτυπη και φαίνεται ότι γίνεται από καπρίτσιο και μόνο. Υπήρξαν αρκετοί ισχυρισμοί ε, και από τον Οργανισμό των Βαλερίδων με πολύ πιο συγκεκριμένα στοιχεία από αυτά που σας δίνω εγώ τώρα. Η διοίκηση στα θέματα αυτά αναγνήρωσε ότι δεν υπήρξαν κάποια κίνητρα ή κάποια αιτιολόγηση για κάποιες νέες τεχνικές εκθέσεις ε, και εμείς έχουμε και μία νομική έκθεση εδώ στα όσα σας παρουσιάζουμε. Δεν έγιναν νέες εκθέσεις και ο ίδιος υπάλληλο που είχε υπογράψει το πρώτο μνημόνιο ε, αμφισβήτησε τις ε, ικανότητες του νομικού ο οποίος αμφισβητούσε την κατάσταση και δημιουργούσε προβλήματα και πρέπει να πω ότι δεν γνωστοποιήθηκε και σε κανέναν. Το θέμα λοιπόν ακολούθησε την πορεία του, εγκρίθηκε το 2019 από την ε, κυβέρνηση των Βελερίδων και ε, εμφανίστηκαν και νέα προστατευόμενα είδη και εξαφανίστηκαν κάποια τα οποία είχαμε στα αρχικά έγγραφα. Ε, και τότε ε, κάναμε σχετικό ερώτημα στα δικαστήρια, το οποίο είναι σε εξέλιξη και παρουσιάσαμε και την σχετική αναφορά ε, εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Με αυτό το αίτημα λοιπόν παρουσιάστηκε και μία έκθεση ενός ανεξάρτητου τεχνικού, περιβαλλοντολόγου και βιολόγου, που έδειχνε για την ορνηθολογική εξέταση που έγινε και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι ανεπαρκή για να ανακηρυχθεί μια περιοχή προστατευόμενη. Θα θέλαμε λοιπόν να καταργηθούν αυτέ οι οποίε περιοχέ οι οποίε ανακαρύχθηκαν ε, έτσι και να γίνουν κατάλληλε βιολογικέ και περιβαλλοντικέ μελέτε για να ξέρουμε αν είναι κατάλληλε για την προστασία των ειδών. Ολοκληρώνω. Μόνο κάτι. Θα μπορούσατε να τα λέτε λίγο πιο αργά, διότι Έχω πέντε λεπτά και πρέπει να τα πω τσίμα τσίμα βγαίνω. Να επαναλάβω κάτι ή να συνεχίσω. Για όλου αυτού του λόγου, ζητάμε λοιπόν από την κυβέρνηση των Βαλερίδων Νήσων να καταργήσει τι περιοχέ που έχει ανακηρύσει και να κάνει τι απαραίτητε βιολογικέ και περιβαλλοντικέ μελέτε, σοβαρέ επιστημονικέ μελέτε, που να δικαιολογούν ότι οι νέε περιοχέ που ανακηρύσσονται ω προστατευόμενε είναι κατάλληλε για τα είδη που θέλουμε να προστατέσουμε. Είναι απλώ μια δικαιολόγητη ε, κίνηση από την αρμόδια διοίκηση. Και ολοκληρώνω λέγοντας, ζητάμε από την Επιτροπή Αναφορών να παραμείνει ανοιχτή αναφορά και να ζητήσουμε από την κυβέρνηση των Βαλερίδων Ίσων όλη την τεχνική και επιστημονική τεκμηρίωση που υπάρχει στο θέμα αυτό, ε, βάσει του οποίου μπορέσαμε να κάνουμε και εμείς την αξιολόγηση ως πληγέντες πολίτες, ε, με τις οποίες αιτιολογούνται αυτές οι νέες περιοχές που θεωρούνται προστατευόμενες. Και ή δυνατόν να κάνετε και μία αποστολή στις Βαλερίδε Νήσες για να δείτε και διεισόμαση την κατάσταση. Θεωρούμε ότι αυτές οι περιοχές ε, περιβαλλοντικές προστασίας πρέπει να αιτιολογούνται καταλήλως με επιστημονική τεκμήριωση. Αλλιώς ε, απατώμαστε ηχτρά και έτσι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ξεκινούμε. Στην Επιτροπή ο λόγος πρώτα. Λουθία Ιγκλέσιας Μπλάνκο. Όχι, Λουίζα Σαμαρέλη, από την ΕΝΒ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Η αναφορά ανατρέχει στον Οκτώβριο του 19. Ακούσαμε το περιεχόμενο από, την, από τον αναφέροντα. Εμείς το καλοκαίρι του 19 με βάση τις πληροφορίες που είχαμε καταλήξαμε ότι δεν υπήρχε καμία αποδεικτική κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι ο ορισμός των προστατευμένων περιοχών δεν πληρούσε τα απαραίτητα κριτήρια. Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να ταξινομήσουν τα, τα πιο κατάλληλα εδάφη ως περιοχές προστασίας των διαφόρων ειδών πτηνών που περιγράφονται στο παράδειγμα 1 και των μεταναστευτικών, των αποδημητικών ειδών. Τα ίδια αυτά μπορούν να είναι και αντικείμενο ειδικών μέτρων προστασία. Το Δικαστήριο της Ένωσης διευκρίνησε ότι τα όρια των ζωνών καθορίζονται μόνο βάσει ονιθολογικών κριτήριων. Δεν υπάρχουν στοιχεία, όπως σας είπα, ότι οι ζώνες αυτές στις Βαλερίδες δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά. Για παραδείγμα, <clears throat> επτά νέες ζώνες είναι σημαντικές για ήδη αετών το πρόγραμμα αποκατάστασης των οποίων χρηματοδοτήθηκε από ένα πρόγραμμα στα πλαίσια του LIFE. Οι αρμόδιες αρχές ε, των Βαλερίδων δεσμεύτηκαν να εντάξουν τις ζώνες αυτές ή να διευρύνουν τις υφιστάμενες στο πλαίσιο του LIFE, του προγράμματος LIFE. Σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες ε, των αναφερόντων για τους, ε, τις επιπτώσεις και τον περιορισμό στην γεωργική και δασική δραστηριότητα, η Επιτροπή καταγράφει ότι ο νόμος που υιοθέτησε η κυβέρνηση για τον ορισμό των περιοχών αυτών δεν περιλαμβάνει περιορισμού στην παραδοσιακή χρήση του εδάφους. Η συμφωνία, το, το κείμενο αυτό, ο νόμος αυτός, ε, απαιτεί τη διατήρηση των ε, αναγκαίων αγροτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή και αναφέρει ότι θα αποφευχθούν περί τι περιορισμοί στην οικονομική, στις τοπικές οικονομικές δραστηριότητε. Η οδηγία οικοτόπων και η οδηγία για τα πτηνά δεν αποκλείουν τη δυνατότητα ανάπτυξη δασικών και γεωργικών δραστηριοτήτων εντός ή γύρω των χώρων προστασίας. Απλώς ζητούν να είναι συμβατές οι δραστηριότητε αυτές με την προστασία των ειδών και των οικοτόπων που έχουν καθοριστεί. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή το, το το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοδότησης της Γεωργίας, μπορεί να συμβάλλει στη χρηματοδότηση μέτρους μέσων συναφών με, την, ε, με δράσεις Natura 2000, όπως δασικής δραστηριότητα και μπορεί να αποζημιώσει την οικονομική ζημία που μπορεί να προκύψει λόγω του ορισμού κάποιας περιοχής ως περιοχής Natura. Η αποζημίωση γίνεται βάσει εθνικών επιλογών για τη χρήση του ΦΕΟΓΑ. Η Επιτοπή γνωρίζει ότι οι Ισπανικές αρχές έστειλαν πληροφορίες για τις νέες ζώνες προστασίας και τη διεύρυνση των δύο υφιστάμενων. Στην τελευταία ενημέρωση του Natura, της βάσης του Natura το Δεκέμβριο του 2019. Τις επόμενες εβδομάδες, το Μάρτιο, θα βγουν τα σχετικά κείμενα στο πλαίσιο του Natura 2000 και θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία αυτά στο κοινό. Χτες λάβαμε μία έκθεση εμπειρογνωμόνων, 100 σελίδες και, δεν τα ξέραμε αυτά, θα τα αναλύσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Θέλουμε να θυμίσουμε ότι οι εθνικές αρχές μπορούν επίσης να αποφασίσουν να ορίσουν συγκεκριμένες περιοχές ως προστατευμένες περιοχές πέραν αυτών που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για να συμπληρώσουν το δίκτυο Natura 2000. Αυτό συμβαίνει συχνά στην Ένωση και υπάρχει πλήρη σχετική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Στρας. Έστρας. Ευχαριστώ. Διαφωνώ με την Επιτροπή. Αυτό που λέει η Επιτροπή είναι ότι η διαδικασία καθορισμού μιας ζώνης είναι σωστή. Ωστόσο, οι ζώνες, ε, οι οκτώ νέες ζώνες στο κέντρο της ε, Μαγιόρκας ε, ορίστηκαν χωρίς να έχουν γίνει τεχνικές επιστημονικές ή ορνηθολογικές μελέτες. Γι' αυτό υπάρχει και μία προσφυγή δικαστική. Διαφωνώ επίσης με την Επιτροπή όταν αναφέρει ότι δεν, δεν, δεν εμποδίζει η γεωργική δραστηριότητα. Ε, αυτό δεν συμβαίνει. Οι νέοι φεύγουν και εγκαταλείπεται η γεωργία. Αυτό λοιπόν είναι σοβαρή βλάβη για τους γεωργούς, για την κτηνοτροφία και για τις δασικές δραστηριότητε, διότι στην ουσία δεν παράγει εισόδημα. Ε, μία ζώνη προστασίας δεν παράγει εισόδημα. Άρα περιορίζεται η οικονομική δραστηριότητα, κάτι που δεν εξηγείται. Θα ζητούσα από την Πρόεδρο το εξή, να μην ανοιχτεί η αναφορά, να ζητήσουμε τις εκθέσεις από τις ε, την τοπική, περιφέρεια από την περιφερειακή μελέτη. Είπε η Επιτροπή ότι πήρε ένα κείμενο 100 σελίδων. Θα την μελετήσουμε κι εμεί. Θα δούμε τα επιχειρήματα. Εμεί δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν επιχειρήματα. Ήταν ένα καπρίτσιο ενός ε, συμβούλου τη περιφερειακή διοίκησης. Πολιτική επιλογή δηλαδή, όχι επιστημονική. Μένει ανοιχτή αναφορά, ζητάμε πληροφορίες και αποφασίζουμε στο μέλλον. Ζητήθηκε αποστολή ε, εκεί από τον αναφέροντα. Ξέρω ότι αποφασίσαμε ήδη, αλλά θα μπορούσαμε ανάλογα με τις πληροφορίες που έχουμε να σκεφτούμε ξανά μία αποστολή εκεί. Είπατε ότι ε, έγινε αποφασίστηκαν οι αποστολές, αλλά οι Βαλεαρίδες είναι ε, μια μεγάλη τουριστική περιοχή που ζει όμως από τη δουλειά των ε, γεωργών. Τα λουλούδια, τα άνθη που βλέπουμε στην ε, Μαγιόρκα. Ας λοιπόν ανοιχτή η αναφορά και θα ζητήσουμε πληροφορίες για να διευκρινίσουμε το ζήτημα και τις μελέτες που απαιτούνται. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλη παρέμβαση. Παρακαλώ κύριε Μαλακόφ. θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζω τη συνάδελφο γιατί έχουμε τα ίδια προβλήματα στη Βουλγαρία με την Natura 2000. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα ε, με τις ΜΚΟ, οι οποίες κάνουν κάποιες προτάσεις, η κυβέρνηση τις εγκρίνει, χωρίς να ε, υπάρχει καμία απολύτως ε, τεκμηρίωση, χωρίς επιχειρήματα. Ε, γι' αυτό ορισμένες ε, περιοχές και πόλεις ε, συμπεριλαμβάνονται στη Natura 2000. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ή με, ποια, με ποιο τρόπο. Απλούστατα επειδή κάποιος αποφασίζει να φτιάξει τα σύνορα αυτών των προστατευόμενων περιοχών χωρίς να έχει απολύτως ιδέα του τι συμβαίνει εκεί. Θα, πιστεύω θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Ωραία λοιπόν. Παρόλο που δεν έχω αρκετές αρμοδιότητες ή πληροφορίες για να προχωρήσω στην αξιολόγηση που μόλις έκανε η Επιτροπή ε, προκειμένου να χαρακτηριστούν κάποιες ε, ζώνες ε, ως προστατευόμενες περιοχές για τα πουλιά. Θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία εδώ. Η αναφέρουσα μας μίλησε για ζώνες που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς ε, σκοπούς ε, ή για το κυνήγι. Άρα λοιπόν ε, θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία γιατί αυτό είναι σημαντικό. Στις ζώνες αυτές συνεπάρχουν διάφορα συμφέροντα. Η Επιτροπή έκανε τη δική της αξιολόγηση και όπως το είπαν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχουν πολλές αποδείξεις στις ζώνες αυτές που συνηγορούν υπέρ ε, του χαρακτηρισμού των περιοχών αυτών ως ζωνών ειδικής προστασίας ε, για πουλιά. Άρα λοιπόν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι δύσκολο να γίνει εμείς ως ε, Επιτροπή ε, λέμε ότι συντρέχουν κάποιοι αποχρόντες ε, επιστημονικοί λόγοι, ούτε ώστε οι ζώνες αυτές να μην χαρακτηρίζονται ως ειδική προστασία. Γι' αυτό θα πρέπει η αναφορά αυτή να παραμείνει ανοιχτή. Ευχαριστώ πολύ. Εάν, επειδή δεν υπάρχει άλλη παρέμβαση θα δώσουμε στον αναφέροντα το λόγο για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να στήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση της τελευταίας ε, πληροφόρησης ε, που σας ε, έδωσα. Τα ορθολογικά κριτήρια είναι τα βασικά. Εγώ θα ήθελα να αξιολογηθούν έτσι όπως ανέκρινε η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων. Ε, υπάρχει ένας ε, τουριστικός οδηγός, δεν υπάρχουν επιστημονικές έρευνες. Αυτό είναι το κείμενο βάσει το οποίο χαρακτηρίζονται αυτές οι περιοχές. Ε, και το πρόγραμμα LIFE δεν ε, αποτελεί μέρος των νέων ζωνών η παραδοσιακή γεωργία γενικά ισοδυναμεί με φτώχεια και επιδοτήσεις. Οι περίφημες ενισχύσεις της ε, Βαλεαρίδες ε, ποτέ δεν χρησιμοποιούνται. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι οι Βαλεαρίδες έχουν αναλογικά περισσότερες ε, ζώνες της Natura 2000 σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση να διευρυνθούν ε, οι ζώνες αυτές γιατί βρισκόμαστε στα όρια. Για να κάνουμε καινούρια πράγματα θα πρέπει να είναι παρκώς τεκμηριωμένα. Αλλιώς η κοινωνία θα δυσπιστεί εναντί της ε, δίκαισης. Γι' αυτό εγώ ζητώ να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, να μελετηθεί το θέμα και να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν τα επαρκή ορνηθολογικά κριτήρια. Εμεί δεν είμαστε κατά του χαρακτηρισμού αυτών των ζωνών, ζωνών προστασία, αλλά εφόσον τεκμηρώνονται επιστημονικά και όχι για ένα καπρίτσιο. Σα ευχαριστούμε πολύ και αφού ακούσαμε τον αναφέροντα, την Επιτροπή και τους συναδέλφους, είναι σαφές ότι ο αναφέρον δεν θέτει να αφιβόλω το ίδιο το μοντέλο χαρακτηρισμού κάποιων ε, ζωνών, αλλά την έλλειψη επιστημονικής ε, τεκμηρίωσης. Άρα προτείνουμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και θα θέλαμε να προτείνουμε εφόσον ε, πήραμε με κάποια καθαίριση έστω τις πληροφορίες αυτές από τον ε, αναφέροντα, γιατί ορισμένες φορές είναι πολύπλεξη διαδικασίε της ε, Ευρωπαϊκή Ένωσης. προκειμένου να φτάσει σε εμά μία πληροφορία την οποία προηγουμένως έχει εξετάσει η Επιτροπή εκ μέρου του αναφέροντα. Έτσι λοιπόν, η δική μας πρόταση θα ήταν να ζητήσουμε πληροφόρηση, περαιτέρω ε, περισσότερες πληροφορίες, γιατί εμείς στο Κοινοβούλιο είμαστε υπέρ της διαφάνειας. Θα ζητούσαμε λοιπόν από την ε, κυβέρνηση ε, τοπική κυβέρνηση των Βαλεαρίδων όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και την τεκμηρίωση στην οποία βασίζει το χαρακτηρισμό της περιοχής αυτής ως προστατευόμενης. Αυτή είναι η πρόταση της Προέδρου. Και στο μέτρο αυτό ευχαριστούμε τον αναφέροντα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Επιτροπή μας είναι η γέφυρα μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών και Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της εμερήσιας διάταξης που είναι το 33 η αναφορά του Ραφαέλ Σάντζεθ Μπογιέρο εξ ονόματος της Αμβίφα για την αποζημίωση στα θύματα της ε, απάτης του φιλατελικού φόρουμ και της αφίνσα. Όπως γνωρίζετε, οι αναφέροντες έχουν πέντε λεπτά για να παρουσιάσουν την αναφορά τους. Θα, παρέμβουν, θα πάρουν το λόγο και δύο ή ο ένας. Και δύο. Ωραία. Αλλά έχετε συνολικά πέντε λεπτά στη διάθεσή της και στη συνέχεια έχετε ε, άλλα δύο λεπτά. Μπορείτε να τα μοιράσετε όπως θέλετε. Αλλά τώρα έχετε συνολικά πέντε λεπτά και στη συνέχεια θα πάρουν το λόγο η Επιτροπή και οι συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι εδώ ενώπιον σας για να σας πω 499.000 Ισπανοί, Πορτογάλοι και Γάλλοι πολίτες ε, πώς η έλλειψη εμπιστοσύνης ε, ε, νιώθουν έναντι στην έλλειψη προστασίας από το Φιλατελικό Φόρουμ και το Αφίνσα. Οι επιχειρήσεις αυτές ε, ξεκίνησαν το 1968 και για περίπου 30 χρόνια λειτουργούσαν χωρίς κανένα πρόβλημα, τηρώντας τις ε, συμβάσεις τους και ασκούντας τη δραστηριότητά τους αγοραπολισίας με νόμιμο και διάφανο τρόπο. Η κατάσταση ήταν γνωστή από όλα τα θεσμικά όργανα της Ισπανίας, την Τράπεζα της Ισπανίας, ε, φορολογικές αρχές και ούτω καθεξής. Ε, τα δημοσίευαν τα στοιχεία τους και εμείς τα πιστεύαμε. Για παράδειγμα, το 2001 δημοσίευση από το Υπουργείο Οικονομίας έλεγε ότι στην Ισπανία η Όμιλος Αφέντσα και το Φιλατελικό Φόρουμ είναι επιχειρήσεις που πάνω από την εγγύηση για εισόδημα είναι και εγγύηση κατά της απάτης. Όλα αυτά άλλαξαν το 9 Μαΐου του 2006 με πολύ διαφορετικό τρόπο. Εκατοντάδες ε, αστυνομικοί ε, με αστυνομικά σκυλιά κλπ. εισέβαλαν σε επιχειρήσεις και όλα αυτά μεταδόθηκαν ζωντανά ε, στην τηλεόραση και τελικά οι εταιρείε χρεοκόπησαν και ρευστοποιήθηκαν τα στοιχεία ενεργητικού τους. Υπάρχει έλλειψη προστασίας και δεν υπήρχε κατάλληλος έλεγχος για τα οικονομικά συμφέροντα των πολιτών. Υπάρχει ο κανονισμός του 2006-2004 ε, και σχετική οδηγία. Επίσης δεν εγκρίθηκαν τα αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά μέτρα για αυτές τις επιχειρήσεις όπως προβλέπει η οδηγία 2005-29 στην αιτιολογική σκέψη 22 όπου ε, ζητά να ε, μην υπάρξουν πολύ μεγαλύτερες απώλειες στους καταναλωτές. Υπάρχει και απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας που θεωρεί ότι η δραστηριότητα της Αφίνσα ήταν ε, ε, μαζική απάτη και ήταν αντίθετη με τα όσα έγιναν μέχρι τώρα. Σύμφωνα με τις απόφαση, οι πελάτες ε, πήγαιναν για να καταθέσουν χρήματα και οι επιχειρήσεις κατα... συμπεριφέροντας σαν τράπεζα. Αυτή η δήλωση έχει άμεσες συνέπειες και οι δύο επιχειρήσεις έπρεπε να ελέγχονται και να εποπτεύονται από τα όργανα ελέγχου της χώρας, σε αυτή την περίπτωση της Τράπεζας της Ισπανίας και εμείς βρεθήκαμε εκτοσημένοι ε, και υπήρχε το άρθρο 19 και η οδηγία του 2004-39 που ε, έδειξαν ότι υπάρχει ε, παράτυπη δραστηριότητα η οποία οδήγησε σε απώλειες στους καταναλωτές. Ε, βρισκόμαστε ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής Αναφορών γιατί θεωρούμε ότι δεν μας προστάτευσαν ως Ευρωπαίους καταναλωτές ένα κράτος μέλος ε, και παρά το γεγονός ότι υπάρχει το άρθρο 69 της ε, Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καθορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα υποπτικά όργανα πρέπει να εγγυώνται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασία στου καταναλωτές και στα οικονομικά του συμφέροντα. Όπως και το άρθρο 1738 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωση, που καθαρίζουν ω θεμελιώδε. δίκαιο την προστασία στο εισόδημα και την ιδιοκτησία και εγγυώνται τη μέγιστη προστασία για τους καταναλωτές. Όλη αυτή η προστασία λοιπόν, η οποία αναφέρεται στα σχετικά άρθρα των οδηγιών και των νομοθετημάτων που αναφέραμε, δεν υπήρξε από την Ισπανική ε, από τις Αρχές ε, και είχαμε μεγάλη ζημία και ατομικά ε, και είναι αποδεδειγμένη. Και φυσικά θα πρέπει οι Ισπανικές αρχές ε, να αναλάβουν τις ευθύνες για τα λάθη που διέπραξαν ε, τα θεσμικά τους όργανα και η μόνη μας ευθύνη είναι ότι εμπιστευθήκαμε αυτά τα όργανα. Όλα τα στοιχεία τα οποία αναφέραμε είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ρύθμιση για αυτές τις επιχειρήσεις και αυτό φυσικά δεν ε, σας απαλλάσσει εσάς από την υποχρέωσή σας ε, να προστατεύετε τους καταναλωτές. Δεν απαλλάσσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν το θεματολόγιο των καταναλωτών να περιλαμβάνει ως βασική αρχή την εφαρμογή της νομοθεσίας, να φροντίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας και να ε, διευκολύνει την αποζημίωση στους καταναλωτές, κάτι το οποίο δεν συνέβη στην περίπτωσή μας. Οι καταναλωτές που εκπροσωπώ εγώ ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει και να παρέμβει προκειμένου να διευκολύνει την αποζημίωση ε, και τον, ε, τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της έλλειψης εφαρμογής της νομοθεσίας και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από τα αρμόδια ισπανικά όργανα και κυρίως από το Υπουργείο Κατανάλωσης να δώσουν στην Επιτροπή Αναφορών όλες τις πληροφορίες για το πώς καταλήξαμε σε αυτή την κατάσταση. Εδώ και 30 χρόνια συνεχιζόταν αυτή η κατάσταση περίπου και το τι σκοπεύουν να κάνουν για να αποζημιώσουν τους 450.000 καταναλωτές ε, που ε, ένα αντικείμενο απάτη εδώ και 14 χρόνια. Υπάρχουν 450.000 καταναλωτέ που παρακολουθούν ε, πολύ προσεκτικά. Μην του απογοητεύσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μιλήσατε 5,5 λεπτά βέβαια. Ε, ένα λεπτάκι λοιπόν παραπάνω. Ναι, θα είμαι σύντομη. Κυρίες και κύριοι, μπορεί να είναι εύκολο να πιστεύετε ότι βρισκόμαστε εμείς εδώ ως ε, μια ίστατη απόπειρα για να ξαναπάρουμε τα χρήματά μας. Ε, δεν θα πρέπει να σας εξαπατά αυτή η απλή τοποθέτηση. Τα τελευταία 14 χρόνια έχουμε ακολουθήσει μια πορεία ε, που φαίνεται ότι προέκυψε από πράγματα τα οποία ήταν επινόηση των αρχών και ένα κράτος το οποίο δεν ρύθμισε τις εσωτερικές του αγοράς. Όλα αυτά ήταν χτυπήματα στην πλάτη ε, απαταιώνων πολιτικών ε, και πραγματικά είχαμε και απόφαση από το ύπατο ανώτατο δικαστήριο το οποίο δεν ε, μπόρεσε να αξιολογήσει τα στοιχεία όπως θα έπρεπε. Κάθε ένα από τα πολιτικά, κυβερνητικά ε, όργανα ή κοινωνικές ε, αρχές τις οποίες αποτανθήκαμε, μας έδωσαν επιχειρήματα τα οποία είναι έολα και δεν ήθελαν να δεχτούν την ευθύνη της Ισπανικού κράτους για αυτό το ατυχές περιστατικό. Γι' αυτό ακριβώ συνεχίζουμε την πορεία μα, ζητάμε διευκρίνηση των γεγονότων, να αναλυφθούν ευθύνε και να υπάρξει αποζημίωση για πράγματα τα οποία δεν έχουμε κάνει εμεί και δεν θα έπρεπε να πληρώσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πληρώσουμε εμεί τη νύφη, διότι αυτοί οι 450.000 άνθρωποι έκαναν επενδύσει και ε, θεμελιώνουν την απόφασή του ε, ακριβώ την εμπιστοσύνη την οποία έδινε η Ισπανική. Ε, χώρα από τις διαφημίσεις, από την ε, δημόσια αναγνώριση και τη θεσμική υποστήριξη. Δεν καλύπτεται λοιπόν η ευθύνη τους ε, από το γεγονός ότι αυτές οι επιχειρήσεις το 2006 και τότε έγινε παρέμβαση χωρίς να υπάρξουν μέτρα εγγυήσεων για τους επενδυτές. Πού ήταν η Τράπεζα της Ισπανίας ε, και οι αρχές οι φορολογικές σε αυτή την περίπτωση. Είναι σαφές ε, ότι δεν εφαρμόστηκε η Ισπανική νομοθεσία και οι ευρωπαϊκές οδηγίες που περιλάμβαναν μια σειρά από εγγυήσει για να μπορέσουμε να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις. Θα θέλαμε να γνωρίζετε ε, ε, ότι όλα αυτά... δημιούργησαν προβλήματα σε οικονομικό επίπεδο, αλλά εμεί δεν είμαστε επενδυτέ ούτε οικονομικοί αναλυτέ. Είμαστε άνθρωποι που χάσαμε τι οικονομίε μα, τι οποίε κάναμε μια ζωή για να τι μαζέψουμε. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Ναι, πολύ σύντομα, δεν έχει μείνει τίποτα. Γι' αυτό ακριβώς κυρίε και κύριοι βρισκόμαστε εδώ έχουμε και προβλήματα υγείας, οικογενειακά προβλήματα και δυστυχώς είχαμε μέχρι και μία αυτοκτονία. Το ε, Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας, στην οποία απευθυνόμαστε, έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσει τα γεγονότα, να υποχρεώσει να διερευνηθούν ε, τα γεγονότα και να υπάρχουν ευθύνες για το κράτος μέλος. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πράγματα για να εγγυηθεί την ισότητα και την προστασία των καταναλωτών σε όλο τον ε, ευρωπαϊκό ενιαίο χώρο. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι γι' αυτό. Η Επιτροπή. Ο κ. Νικές Σατώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε την θέση μας μετά από μια σειρά αναφορών τις οποίες συμβάλαμε. Το επιπρόσθετο υλικό που αναφέρεται υπογραμμίζει ότι το ποινικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ε, Ισπανίας θεωρεί ότι η εταιρεία κάνει οικονομική δραστηριότητα και καταλήγεται ότι αυτό σημαίνει πως ε, υπάγεται στην ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική νομοθεσία η δραστηριότητα αυτή. Ωστόσο, όπω είπαμε σε προηγούμενε απαντήσει μα, οι δραστηριότητε τη Φιλατέλικο και τη Αφίνσα δεν είχαν εξουσιοδοτηθεί από την Εθνική Υπηρεσία ε, ε, Χρηματιστηριακών Αξιών και άρα δεν υπάγονται στις δραστηριότητε τη υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ιδίω για την εμπορία χρηματοοικονομικών μέσων και την πρόθεση στην αγορά, το MIFID. Η απόφαση του 2017 δεν αλλάζει το συμπέρασμα αυτό, γιατί οι, υπο, οι προϋποθέσεις στο MIFID δεν αλλάζουν. Εξού και η οδηγία, η οδηγία αυτή καλύπτει πιστοτικά ιδρύματα που είναι εποπτευόμενα ιδρύματα και παρέχουν υπηρεσίες όπως ε, εκτέλεση εντολών των πολιτών, παραλαβή και μεταβίβαση εντολών, επενδύσεις και διαχείριση χαρτοφυλακίου. Για να υπαχθεί μια υπηρεσία στι επενδυτικέ δραστηριότητε, μια, μια δραστηριότητα θα πρέπει να σχετίζεται με χρηματοοικονομικά εργαλεία, ομόλογα κλπ. Η οδηγία έχει ρητή και αποκλειστική λίστα τέτοιων Ινστιτούτων στο παράδειγμα 1 τμήμα Γ η συμπεριφορά δραστηριοτήτων που και τη συγκεκριμένη δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών. Οι συγκεκριμένες δράσεις της αναφοράς δεν υπάγονται σε αυτά και δεν λαμβάνουν την προστασία της οδηγίας στους αγοραστές και πολιτές των προϊόντων αυτών. Οι οδηγίες για το πρόγραμμα αποζημίωσης των επενδυτών που προβλέπει την αποζημίωση ε, σε περιπτώσεις ε, απώλειας ε, ενεργητικού δεν εφαρμόζεται κατά συνέπεια. Σε ό,τι αφορά τις ατασταλίες που περιγράφεται στις Ισπανικές Αρχές και στη δικαστική διαδικασία έναντι των δύο αυτών εταιριών και τις αντιφάσεις που πιθανόν υπάρχουν σε αποφάσεις των δικαστηρίων είναι ζητήματα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής, είναι εκτός της δικής μας αρμοδιότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Σταράς, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τους αναφέροντες, την ε, Ένωση Θυμάτων του Φόρουμ Φιλατέλικο και της Αφίντσα. Είπαν και σωστά ότι εκφράζουν χιλιάδες ανθρώπους που κατεύθυνσαν τα χρήματά τους στις δύο επιχειρήσεις, το Φόρουμ Φιλατέλικο και την Αφίνσα, που ήταν εξειδίκευση στο εμπόριο γραμματοσύμων. Είναι εδώ διότι η αναφορά τους, η Επιτροπή Αναφορών μάλλον, είναι η Επιτροπή που είναι πιο κοντά στον πολίτη, όπου ο πολίτης ελπίζει να βρει μια λύση στην προστασία των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων πέρασαν ένα γολγοθά δικαστικό. Αντιφατικές αποφάσεις μεταξύ του ανώτατου δικαστηρίου και του ποινικού τμήματος του δικαστηρίου. Πολλά άτομα επλήγησαν στην υγεία τους, ψυχολογικά αισθάνθηκαν ότι τα δικαιώματά τους καταπατούνται και ήρθαν εδώ να ζητήσουν από εμά να κάνουμε κάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε. Η Επιτροπή είναι όργανο πίεσης και σκέψης. Δεν είναι δεσμευτικό όργανο, σε πολλές περιπτώσεις όμως πρέπει να, να κάνουμε τα κρατημένη να σκέφτονται. Ζητώ λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να στραφούμε προς τις ισπανικές αρχές για να δούμε πώς οι αναφέροντες θα μπορούσαν να αποζημιωθούν ως καταναλωτές εκεί όπου η ένομη τάξη και το κράτος απέτυχαν. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να τους δώσουμε μια διέξοδο, να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να ζητήσουμε από τις Ισπανικές Αρχές να σκεφτούν πώς θα μπορέσουν να αποζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί ως καταναλωτές. Ευχαριστώ. Μπούσμαν. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε επίσης και τους αναφέροντες για την αναφορά αυτή. Εγώ εδώ είμαι κατά εντολή του συναδέλφου Ρεαρέγκο ο οποίος θέλει να πάρει το λόγο. Οι δικές μου ε, πληροφορίες αφορούν χιλιάδες ε, Ευρωπαίων πολιτών οι οποίοι επένδυσαν τα χρήματά τους στο, ε, ε, στο φιλατελικό φόρουμ ε, βάσει ένα συστήματος πυραμίδων. Ε, όπως είπαμε, έκλεισαν. Έκλεισε η επιχείρηση αυτή από την Ισπανική αστυνομία. Ε, χιλιάδες είναι οι πληγέντες επενδυτές και είναι δικαιολογημένα τα αιτήματα αποζημίωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιληφθεί της υπόθεση αυτής και σας παρακαλώ η αναφορά αυτή να παραμείνει ανοιχτή. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κάνιας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Οι πολίτες ε, Ε, εκχωρούν στη διοίκηση τον έλεγχο, τη ρύθμιση και την ε, εποπτεία των δραστηριοτήτων τους ως ε, πολιτών. Και δυστυχώς η περίπτωση αυτή, αυτού του φαινομένου πυραμίδας, που κατέστρεψε χιλιάδες πολιτών και τους έβαλε σε ολέθριες προσωπικές καταστάσεις. θυμάμαι τέτοιες περιπτώσεις ε, σε μια ε, συγκέντρωση που είχε γίνει στη Βαρκελόνη από θύματα αυτής της υπόθεσης. Ε, θα πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν μια επιχείρηση εμπορευματοποιεί κάτι το οποίο είναι εκτός όπως είναι τα γραμματόσημα ε, δεν ήταν ε, μια, ένα φαινόμενο πυραμίδα το οποίο κινείται σε μυστικούς ε, κύκλους. Όχι, ήταν το φιλατελικό φόρουμ. Και ορισμένοι κυβερνητικοί κύκλοι συμμετείχαν σε κάποιες τέτοιες πράξεις. Αλλά όταν έκρισε το πρόβλημα είπαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό γιατί ήταν εκτός του δικού τους ελέγχου. Δεν εμπίπτει στη δική τους εποπτεία. Ε, τι μπορεί να γίνει, είτε να μην γίνει τίποτα, αυτό το οποίο έγινε, ή γιατί ε, θυμάμαι ότι στην Ισπανία και σε άλλες ευρωπαϊκές ε, χώρες 700 εκατομμύρια ευρώ αφιερώθηκαν στην διάσωση ε, επιχειρήσεων προκειμένου ε, να γίνουν κάποιες ε, στις οποίες είχαν γίνει επενδύσεις υψηλού κινδύνου. για τέτοιες δραστηριότητες οι οποίες επίσης ήταν εκτός αρμοδιότητας του εποπτείας. Ε, άρα λοιπόν οι τράπεζες είχαν αυτή την κάλυψη ενώ οι ιδιώτες δεν την, έχαν, δεν την έχουν γιατί ε, πρόκειται για τα τεράστια ποσά όπως σας είπα Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι αφορά να γίνει μια, ε, θα πρέπει να γίνει μια σαφής διάκριση μεταξύ της υποχρέωσης του κράτους και της ε, ευθύνης του κράτους. Και στην περίπτωση αυτή έχουμε, θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Ο κύριος Λαμπακόφ. Ευχαριστώ. Ε, συμφωνώ απολύτως με τους προλαλήσαντες. Θα ήθελα απλώς να προσθέσω ότι πρόκειται, για 450.000 ε, άτομα στην Γαλλία και στην Ισπανία εδώ που είναι θύματα. Δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί ε, βρίσκονται ε, και βρίσκονται εδώ μόνο για να πάρουν τα χρήματά τους, αλλά γιατί επιθυμούν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και θεωρώ ότι το Ισπανικό κράτος έκανε έκδηλα ε, σφάλματα, γιατί είναι αδύνατο να δρουν ε, τέτοιες επιχειρήσεις απουσία ελέγχων. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθούν κάποιοι τρόποι αποζημίωσης των ανθρώπων αυτών, τουλάχιστον ε, ε, όσον αφορά τα όσα προβλέπονται από τις, ε, από τις συμβάσεις που έχουν κάνει, τα συμβόλαια. Βεβαίως η αναφορά αυτή θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Ο κύριος Σαλίμπα. Εδώ είμαστε μάρτυρες μιας Ε, ε, ε Υπάρχουν ε, ευάλωτες ομάδες καταναλωτών στην αγορά μας, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υιοθετήσει κάποιες νομοθετές διατάξεις προκειμένου να προστατευθούν οι καταναλωτές. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι σε τέτοιες ε, περιπτώσεις είναι οι οικονομίες ζωής ε, που επενδύουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ισπανία, αλλά είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε χώρες όπου εκατοντάδες άνθρωποι ε, επενδύουν ολόκληρες τις οικονομίες τους κάπου, σε κάποια σχήματα. Και ε, νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή υπάρχουν ε, ζητήματα τα οποία δεν έχουν διαλευκανθεί πλήρως. Γι' αυτό θα πρέπει η αναφορά αυτή να παραμείνει ανοιχτή, ούτω ώστε να έχουμε περισσότερα στοιχεία και προκειμένου να απαιτήσουμε να υπάρξει καλύτερη προστασία των καταναλωτών. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Ασμακοπούλου. Um, Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή ε, βεβαίως ε, καταλαβαίνω, κατανοώ τα νομικά επιχειρήματα τα οποία ε, προβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, εμείς ως μέλη της ε, Επιτροπής εδώ και ως ε, πολιτικοί έχουμε μια πολιτική υποχρέωση, ακόμα και μια ηθική υποχρέωση ε, υπό το πρίσμα των διαστάσεων της ζημίας που έχει, που έχει γίνει. Και οι λογικές προσδοκίε που έχουν οι άνθρωποι αυτοί ότι θα έπρεπε να προστατευθούν, ότι θα προστατεύονται ε, και θα είχαν μια ευρωπαϊκή κάλυψη. Αυτό καθιστά αναγκαίο να εξετάσουμε την κατάσταση αυτή με τον πιο, ή δυνατόν με πιο εξαναλυτικό τρόπο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε σαφώς περισσότερες πληροφορίες και περισσότερες ε, λεπτομέρειες και στη δική μου χώρα υπάρχουν παρόμοιες καταστάσεις, οι οποίες ε, ε, έπληξαν ε, πολλές οικογένειες, πολλούς πολίτες. Ακούσαμε τι έγινε στην Ισπανία και νομίζω ότι για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει η αναφορά αυτή να παραμείνει ανοιχτή. Ευχαριστώ. Ο αναφέρον τώρα έχει δύο λεπτά για να κλείσει την αναφορά. Ευχαριστώ. Καταρχάς ε, θα ήθελα να πω στην ε, τελευταία ομιλητρία που μας υποστήριξε εμείς είμαστε διατεθειμένοι να σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, οτιδήποτε χρειάζεται τα διαθέτουμε και μπορούμε να σας τα δώσουμε. Κάτι άλλο, αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς δεν θεωρούμε ότι η επιχείρηση αυτή ε, δεν θα έπρεπε να ελέγχεται από την οδηγία MIFID, από τον τρόπο με τον οποίο ήταν ε, η σύσταση τη Έπρεπε η Τράπεζα της Ισπανίας να υποχρεούται να ελέγξει αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν είναι ε, η προϊόν επενδύσεων, αλλά σύμφωνα με την απόφαση έπαιρναν χρήματα που ήταν καταθέσεις ε, προθεσμιακές και ε, χρόνο θα έπρεπε απλώ να έχουν κάποια επιτόκια. Ε, λειτουργούσαν λοιπόν σαν κανονικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, σαν τράπεζα και ε, θα έπρεπε λοιπόν να ελέγχεται από τη τράπεζα της Ισπανίας ε, ή να το κλείσουν. Ε, από την πρώτη στιγμή όμως, όχι να περιμένουν 30 χρόνια. 30 χρόνια, όπως έλεγε ο κύριος Κάνιας, όλα τα όργανα της Ισπανίας, όλα σε εξουσίες, η εκτελαστική, η δικαστική, συμφωνούσαν ότι είναι πάρα πολύ καλή η λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ε, νομίζω ότι πρέπει να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας και πραγματικά ε, θα κάνετε πολύ χαρούμενους 450.000 ε, ανθρώπους αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ τους αναφέροντες που ήταν εδώ σήμερα μαζί μας. Ε, μετά από τα όσα ακούσαμε από τους αναφέροντες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα μέλη της Επιτροπής, η πρόταση της Προεδρίας είναι να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και μετά από τις ε, παρατηρήσεις ε, και τα σχόλια των ε, μελών από όλε τις κοινοβουλευτικές ομάδες θα προτείνουμε να αποστείλουμε και επιστολή στις Ισπανικές Αρχές προκειμένου να πιέσουν και να δούμε πώς μπορούμε να ε, επανορθώσουμε αυτή τη ε, μεγάλη ζημιά που έπληξε τόσες χιλιάδες ε, Ισπανούς, Πορτογάλους και Γάλλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους αναφέροντες που ήταν εδώ σήμερα το απόγευμα. Συνεχίζουμε τώρα, σημείο 34 της ημερήσιας διάταξης, αναφορά 939 του 2018 από τον Αντρέι Χαλίσκι από την Πολωνία για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα ε, Χρηστής ε, ε, Διοικητικής Συμπεριφοράς. Δεν είναι εδώ αναφέρω. Να δώσω το λόγο στην Επιτροπή, στην κυρία Κρίστενσεν. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο για την αναφορά αυτή. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο κύριος Χαρίτσκι ζητά ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Καλής Διοικητικής Συμπεριφοράς ή κάποια τέτοια πρότυπα να περάσουν ως οδηγία ή ως κανονισμός για να υποχρώνουν τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν τις σωστές διοικητικές πρακτικές. Η Επιτροπή αναγνωρίζει βεβαίως την σημασία της χρηστής διοίκησης και έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει τις αρχές χρηστής διοίκησης σε όλες τις επαφές της με το κοινό. Όπως και τα άλλα όργανα της Ένωσης, η Επιτροπή το 2000 υιοθέτησε το δικό της κώδικα χρηστής διοίκησης και καλής διοικητικής συμπεριφοράς στις σχέσεις της με το κοινό. Είναι ένας γενικός κώδικας που εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους όπου δεν υπάρχει ειδικό κανόνικος κώδικας. Οι αρχέ του κώδικα υλοποιούνται σε καθημερινή βάση και η Επιτροπή τηρεί την υποχρέωσή της να εξυπηρετεί το ευρωπαϊκό κοινό. Κάποιες από τις αρχές αυτές σα είναι γνωστές. Νομιμότητα, αναλογικότητα, δικαίωμα αρχή ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένε διαστάσεις των διοικητικών διαδικασιών όπως ε, χρηματοοικονομική διαχείριση, πρόσβαση σε έγγραφα, προστασία δεδομένων, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί που περιγράφουν τα ουσιαστικά και δικονομικά δικαιώματα των πολιτών έναντι των οργάνων της Ένωσης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι αυτοί οι κανόνες αφορούν μόνο την ευρωπαϊκή διοίκηση η διοργάνωση της εθνικής διοίκησης δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες της Ένωσης. Δεν υπάρχει νομική βάση στη συνθήκη για να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν πρότυπα οθής διοικητικής συμπεριφοράς σε εθνικό επίπεδο. Θυμίζω λοιπόν ότι το άρθρο 197 της συνθήκης αναφέρεται στην πιθανότητα για την Ένωση να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών για την βελτίωση της διοικητικής τους ικανότητας. Υπογραμμίζω ωστόσο εκ νέου ότι δεν υπάρχει υποχρέωση των κρατών μελών να χρησιμοποιήσουν την δυνατότητα αυτή. Και ούτως ή άλλως δεν υπάρχει συνθήκη καμία, κανένα άνθρωπο να προβλέπει εναρμόνιση μόνο τη διοικητική ικανότητα καλύπτει. Συμπερασματικά, η άποψη επιτοπής είναι ότι η Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα να δράσει, όπως μας ζητά ο αναφέρον. Thank you, Chair. I uh, tend to agree with the assessment of the of the committee. Κύριος Βίνσεν, συμφωνώ. Η δέουσα η χρηστή η διοικητική πρακτική σε όλα τα κρατη είναι στόχος όλων και ένας μεγάλος στόχος και για τους πολίτες και για την καλή διακυβέρνηση. Το να καταστήσουμε κάτι τέτοιο υποχρεωτικό για τα κράτη-μέλη είναι εκτός της συνθήκης. Συμφωνώ λοιπόν ότι το ότι δεν υπάρχει νομική βάση στη συνθήκη για την εφαρμογή από την Ευρώπη, την επιβολή την Ευρώπη κανόνων στην εθνική διοίκηση. Το ζήτημα αυτό μπορούμε να το θέσουμε και σαν μια προσπάθεια βελτίωσης μας ένα καλό πρόγραμμα που μπορεί να αναπτυχθεί, αλλά το να υιοθετήσουμε κάτι το υποχρεωτικό, οδηγία ή κανονισμό, είναι αδύνατο. Καλό θα ήταν για τους πολίτες και λυπάμαι που λείπει ο κύριος Χαλίτσκι για να υποστηρίξει την αναφορά του, αλλά θα ήταν μια καλή απόφαση να προσπαθήσουμε να ενημερώνουμε ο ένας τον άλλον για τις καλές πρακτικές μέσω της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Είναι λίγο προβληματικό. Ξέρουμε τι είναι η χρηστή διοίκηση. Πάει παραπέρα από αυτό που είπατε εδώ. Το έχουμε στην Δανία. Δεν το σέβονται πάντα, αλλά υπάρχει στη διοίκηση που είναι η αρχή της υπηρεσίας. Δηλαδή, για να το εξηγήσω, ο πολίτης είναι στο κέντρο. Τίποτα δεν υπάρχει που προστατεύει τους πολίτες. Ο στόχος είναι η προστασία των πολιτών, όχι των υπαλλήλων. Εμείς για χρόνια ζητούσαμε κάτι τέτοιο στην ετήσια έκθεση του διαμεσολαβητή και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί. Όχι μόνο καλά λόγια. Κάπου στο χάρτη υπάρχει μία παράγραφος. Ξέρω ότι η παράγραφο, ότι ο χάρτης εφαρμόζεται μόνο για την Ένωση, δεν εφαρμόζεται τα κράτη-μέλη, είναι παράξενο. Έχουμε διαμεσολαβητή στην Ένωση και πρέπει να ζητήσουμε να υπάρξει νομοθεσία στην Ένωση. Αλλά βλέπετε πόσο δύσκολο είναι να εφαρμόσουμε και άλλους κανόνες που υπάρχουν. Ας πούμε πρόσβαση στα έγγραφα. Πιστεύω ότι πρέπει να πάμε παραπέρα. Δεν αρκεί να δακρύζουμε γιατί δεν έχουμε νομική βάση. Όλοι ξέρουμε ότι αν περάσουμε στη διοίκησή μας, στο εθνικό επίπεδο, την αρχή της ε, υπηρεσίας προς τον πολίτη, θα σώσουμε πολλά πράγματα. Και να πούμε στα κρατημέλη, γιατί να μην το κάνουμε. Όλο ένα και περισσότερο ακούω ότι δεν υπάρχει πλήρη διαφάνεια γιατί πρέπει να προστατεύσουμε και τον υπάλληλο. Λάθο! Από τη στιγμή που υπάρχουν μέτρα προστασίας του υπαλλήλου δεν προστατεύεται ο πολίτης. Δεν είμαι ικανοποιημένη από την απάντηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα για να δημιουργήσουμε σωστή, χρηστή διοίκηση με τον πολίτη στο κέντρο. Και θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε, να χρησιμοποιηθεί εκείνη η παράγραφος στο χάρτη και να πούμε να ξεκινήσουμε από εδώ, στην Ένωση. Ο διαμεσολαβητής είχε παρουσιάσει κάτι καθηγητήριες γραμμές. Για την Ένωση και να δώσουμε εκεί την έμφαση. Γιατί όλοι θα κερδίσουν νομίζω. Και να το συζητήσουμε και με την ε, Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Τι να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Οι σοσιαλιστές ε, είμαστε βεβαίως ε, πλήρως σύμφωνοι ο κώδικας της ε, δεοντολογικής συμπεριφοράς των δημοσίων επαλλήλων να περιλαμβάνει τα, τους υπαλλήλου της διοίκησης, γιατί η νομοθεσία αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες μέλη. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα ως Ευρωπαϊκή Ένωση η εφαρμογή ενός τέτοιου δοντολογικού κώδικα. Αλλά είναι βεβαίω σημαντικό να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Αν εμείς ως Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο δεν εφαρμόσουμε οι ίδιοι το πιο υψηλό, δυνατό επίπεδο υποχρεώσεων σε σχέση με τον κώδικα αυτό, τότε, μόνο τότε θα δώσουμε ένα βέλτιστο παράδειγμα το οποίο μπορεί να ακολουθεί από τις χώρες μέλη. Την τελευταία εβδομάδα η έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή υιοθετήθηκε για την προηγούμενη χρονιά και ήταν σημαντικό ο κώδικας αυτός να αποβεί ε, δεσμευτικός, υποχρεωτικός δηλαδή. Ωραία λοιπόν, προτείνουμε ο κώδικας αυτός να ε, βασιστεί σε ισχυρά εθνικά στοιχεία και ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να μπορεί να συνεχίσει να ασκεί πίεση προς χώρες μέλη. Είμαστε υπέρ του να μείνει συνεπώς ανοιχτή η αναφορά αυτή. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Η αρχική μου πρόταση ήταν να κλείσει, αλλά το να επιμείνουμε στην Επιτροπή και τον αρμόδιο επίτροπο, ο οποίος θα έρθει εδώ το Μάρτιο, προκειμένου να δώσει μια απάντηση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, γιατί ε, δεν θεμελιώνεται μένει στις συνθήκες, αλλά θα πρέπει να συνεχίσει η συνεργασία ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον αρμόδιο επίτροπο κ. Σέσκοβιτς. Ε, πρέπει να διατυπώσουμε αυτή την ε, πρόταση. Δεν ξέρω, συμφωνείτε, κύριε Όγκεν. Ε, ναι, ευχαριστώ, αλλά θα πρέπει να προσκληθεί και ο διαμεσολαβητής στην Επιτροπή προκειμένου να δούμε πώς θα εφαρμοστεί στο ευρωπαϊκό σύστημα. Ε, θα ήταν ο πιο γρήγορος τρόπος. Άρα λοιπόν η πρόταση ήταν να κλείσει, αλλά να το ανοίξουμε προς τον αρμόδιο επίτροπο και ε, τον διαμεσολαβητή. Και τώρα θα περάσουμε στο τελευταίο σημείο ε, που αφορά την αναφορά του Περ Πάολο Βόλπε που αφορά για την ε, διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής ως ε, ελεγκτικού οργάνου. Ε, Παρίσταται εδώ οι αναφέροντες, γι' αυτό τους καλωσορίζω. Έχετε πέντε λεπτά για να εξηγήσετε την αναφορά σας. Στη συνέχεια θα πάρει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε τη δυνατότητα να συζητήσω δημοσίω την αναφορά μου για τη διακριτική εξουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εποπτεία για την εφαρμογή του δικαίου τη Ένωσης εκ μέρου των κρατών μελών. Η ανάγκη να υποβάλουμε αυτή την αναφορά ε, προκύπτει από το μεγάλο περιθώριο ε, το οποίο δίνεται από τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το αν και κατά πόσο θα ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώπιον των κρατών μελών όταν βρισκόμαστε ε, σαφώς μπροστά σε μια κατάφορη παραβίαση των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει τόσο ευρύ ε, ε, περιθώριο και τόσο μεγάλη διακριτική ευχέρεια για να νομοθετήσει και να υποβάλει προτάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο την τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας ε, και την νομολογία ε, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν υπάρχει παραβίαση του δικαίου της Ένωσης από πλευράς κράτους μέλους θα πρέπει πάντα και να παρεμβαίνει ξεκινώντας μια διαδικασία επιπαραβάση σε συγκεκριμένους και σαφείς χρόνους ε, για να επιτρέψει σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τα οποία φυσικά έχουν και συνέπειες στη ζωή και τα δικαιώματα των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κάποια αδράνεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να απαντήσει ε, σε θέματα προϋπολογισμού ή κρατικές ενισχύσεις. Απ' την άλλη όμως είναι και επιπολαιότητα και καθυστέρηση των καταγγελιών των ε, πολιτών οι οποίες γίνονται γιατί υπάρχει παραβίαση των θεμελιών δικαιωμάτων που έχουν αντίκτυπο για χιλιάδες πολίτες και εργαζομένους και για τις οικογένειές τους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το γεγονός ότι αδιαφορεί έτσι ε, σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο κόστος για τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, τηρεί το ρόλο της ως θεματοφύλακα των συνθεκών και ορισμένες φορές και τον διαγράφει και επομένως ε, είναι και άχρηστη η διαδικασία επιπαραβάση ε, και το γεγονός ότι είναι στη διακριτική ευχαίρεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδηγεί σε έλλειψη εμπιστοσύνη των, των πολιτών ενώπιον του Θεσπικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία κανονικά θα έπρεπε, συγγνώμη, ε, αν μπορείτε σας παρακαλώ λίγο πιο αργά. Είναι και τέλος της ημέρας, ε, εκεί είμαστε όλοι κουρασμένοι οι οποίοι έχουν καθήκον να εποπτεύουν για το σεβασμό των δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας δώσω ένα προφανές παράδειγμα της αδράνειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο είχε συνέπειες για τη ζωή των ανθρώπων. Να αναφέρουμε το θέμα που αφορά την ε, παραβίαση των ε, συμβάσεων ορισμένου χρόνου και τη διαδικασία επιπαραβάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και τις τρεις έρευνες οι οποίες είναι ανοιχτέ από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σε θέματα διαχείρισης. Σας παρακαλώ λίγο πιο αργά, κύριε Βόλπε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ε, ε, απαντήσεις της ε, στους πολίτες που καταγγέλουν τη συμπεριφορά αυτή, απαντούν ότι δεν μπορούν να ε, χρησιμοποιήσουν τη διαδικασία επί παραβάση και επομένω οι πολίτε θα πρέπει να αποτανθούν στι εθνικέ αρχέ. Η ε, δήλωση αυτή είναι αληθή μόνο εν μέρη. Ναι, στι περισσότερε περιπτώσει, τα εθνικά δικαστήρια πρέπει ε, να απαντήσουν, αλλά ουσιαστικά είναι αυτά τα οποία παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο και όσον αφορά τη συμβάση ορισμένου χρόνου στην Ιταλία η διαδικασία επί παραβάση για τα Ιταλικά δημόσια σχολεία και την κατάχρηση αυτών των βάσεων ορισμένου χρόνου. Έκλεισε πάρα πολύ γρήγορα και υπήρχε μια νέα διαδικασία επί παραβάση για όλο το δημόσιο τομέα και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και μετά από έξι χρόνια είχαμε και την επιστολή τη σχετική και ε, παρόλα αυτά οι Ιταλικές αρχές ε, παραβιάζουν την οδηγία 9970. Η έναρξη μια διαδικασία επιπαραβάση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει έμεσε συνέπειε για τι μεμονωμένε περιπτώσει. Διότι το να ε, τηρεί ένα κράτο μέλο ε, το κοινοτικό δίκαιο λύνει και το πρόβλημα του μεμονωμένου πολίτη. Μια και τα δικαστήρια τα ίδια είναι αυτά τα οποία δεν συμμορφούνται με το δίκαιο τη Ένωση. Είναι η περίπτωση που συζητήθηκε ήδη στην Επιτροπή των Αναφορών του αρμοδίου δικαστή που ήταν αυτό ο οποίο δεν συμμορφώθηκε στο δίκαιο τη Ένωση, παρά το γεγονό ότι υπήρχε σε εξέλιξη μια διαδικασία επί παραβάση. Ζητάμε λοιπόν αποφασιστική παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να υποχρεώσει με όλα τα μέσα, ακόμα και με τροποποίηση των κανόνων ή και των συνθήκων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποχρεούται να ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση όταν έχουμε παραβίαση του δικαίου τη Ένωση από πλευρά κράτου μέλου και έτσι δεν θα υπάρχει διακριτική ευχαίρεια από πλευράς Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αν και κατά πόσο θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση, η οποία κινεί βάρο και των οικογενειών και των πολιτών. Ευχαριστώ, κύριε Βόλυπε. Η Κομισιόν, η ο κύριος William Sleeth. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που επιτρέπετε να συμπληρώσουμε τα γραπτά σχόλια της Επιτροπής. Καταρχάς, όπως τονίζει και ο αναφέρον, ο τομέας αυτός είναι καθοριστικό, καθοριστικός. Ο ρόλος της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των συνθήκων είναι ουσιαστικός και η πρόεδρος κυρία Βαντελάιν τόνισε ότι η εφαρμογή της κοινωτικής νομοθεσίας είναι προτεραιότητα της νέας Επιτροπής. Επίσης, καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζουν και οι καταγγελίες των ατόμων αλλά και αναφορές για να γνωρίσουν στην Επιτροπή πιθανές παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και συχνά αποτελούν το ξεκίνημα μιας διαδικασίας παραπομπής. Η αξία δεν αγνοείται. Η Επιτροπή εξετάζει προσεκτικά κάθε ατομική καταγγελία. Ωστόσο, οι διαδικασίες παραπομπής και η επιδίωξη ατομικής αποκατάστασης είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι. Όπως γνωρίζετε καλά, η διαδικασία παραπομπής δεν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση ενός ατόμου ή να επιτρέψει μια ατομική αποκατάσταση, αλλά είναι ένας διάλογος αν χρειαστεί, και ή αν χρειαστεί εθνική, όχι ατομική, αποκατάσταση της ζημίας μεταξύ Επιτροπής και κράτους μέλους. Η εθνική νομοθεσία είναι αυτή που αντιμετωπίζει ατομικά αιτήματα αποζημίωσης και η αποκατάσταση καλύτερα να ζητείτε όσο πιο κοντά στον πολίτη γίνεται. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε πώς έχει κατάσταση τη διαδικασία παραπομπής. είναι ουσιαστικό η Επιτροπή να έχει ελευθερία και διακριτική μεταχείριση στον τρόπο με τον διακριτική, το δικαίωμα να διακρίνει στον τρόπο με τον οποίο προχωρεί στην παραπομπή. Ο στόχος είναι να υπάρξει συμμόρφωση του κράτους μέλους με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να πάψει το συντομότερο δυνατό η παραβίαση της νομοθεσίας. Δεν μπορεί με τον ίδιο τρόπο να αντιμετωπιστούν όλες οι παραπομπές. Δεν εξυπηρετεί. Η Επιτροπή ήταν ξεκάθαρη στην ανάγκη να υπάρξει προτεραιοποίηση. Στην ανακοίνωσή της το 2016 είχε θέσει μια στρατηγική προσέγγιση εφαρμογής της κοινοτικής πολιτικής με στόχο την αντιμετώπιση των σημαντικότερων παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Πιστεύουμε ότι η προτεραιοποίηση είναι βασική σημασία διότι δίνει έμφαση στις διαφορετικές παραβιάσεις του δικαίου, εκείνες δηλαδή που βλάπτουν σημαντικότερα τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτό είναι το πλεονέκτημα πρόοδου σε συγκεκριμένους τομείς, π.χ. το περιβάλλον. Οι καταγγελίες και αναφορές λοιπόν είναι ουσιαστικό στοιχείο του συστήματος της Ένωσης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Η Επιτροπή σε κάθε περίπτωση όταν δεν θέλει να προχωρήσει σε παραπομπή, εξετάζει τον καλύτερο μηχανισμό επίλυσης του προβλήματος και θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε το ενδεχόμενο αυτό όταν υπάρχουν αναφορές για τις περιπτώσεις εκείνες που θεωρούμε πιο κρίσιμες. Προσοχή, το ότι έχουμε δικαίωμα δεν σημαίνει ότι έχουμε αυθαίρετο δικαίωμα να επιλέγουμε την διαδικασία. Πρέπει να εξηγούμε. Και αυτό το έχει πει ακριβώς και το Δικαστήριο της Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε εξαντλήσει το κατάλογο των ομιλητών. Κυρία Σάουκεν. Έχετε δίκιο. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η τάση το να αφήσουμε στα εθνικά δικαστήρια αυτή τη δουλειά και αυτό είναι, ε, αυτή είναι η συνήθις πρακτική και μάλιστα ε, επιδεινούνται ε, όσο βρίσκομαι εδώ και βάζουμε πολύ βαρύ φορτίο στις πλάτες των πολιτών. σε ορισμένε χώρε δεν είμαστε εξαντλημένοι, εξουθενωμένοι για λόγου οικονομικού, έλλειψη χρόνου κλπ. Αλλά σε άλλε χώρε ε, δεν είναι δυνατόν να πούμε, να πόκιτε σε εσά να λύσετε το πρόβλημα. Εμείς έχουμε εκδώσει ένα κώδικα διοντολογίε ε, και σε εσά ε, απομένει να τον εφαρμόσετε. Ε, θα πρέπει να πάρουμε, πάρει η Επιτροπή πολύ πιο σοβαρά την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ε, πολλές φορές βλέπουμε δεν σημαίνει τίποτα γιατί οι πολίτες δεν έχουν ε, την ε, εξουσία ακόμα και στη δική μου χώρα την Δανία ε, τα πράγματα μπορούν να λυθούν μόνο με ε, συζήτηση, με διάλογο, γιατί υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα. Ε, υπάρχουν μάλλον λόμπι που εκείνες έχουν την εξουσία για να περάσουν τις δικές τους, τα δικά τους συμφέροντα. Σε πολλές χώρες γίνονται πολλαπλές εφές και τελικά οι πολίτες εγκαταλείπουν ε, θα πρέπει να υπάρξει ένας σεβασμός για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι σημαντικό η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει το ρόλο της ε, σοβαρά. Και νομίζω ότι το άρθρο 265 της Συνθήκης το καθιστά σαφές. Γιατί λέμε ότι αν δεν ε, όταν πρέπει η Επιτροπή να παρέμβει στην ε, περίπτωση αποτυχίας. Ε, δεν ταιριάζει αυτή η συνταγή σε όλους. Δεν γίνεται να, να εγκαταλείψουμε τα πάντα στην αρμοδιότητα των χωρών μελών. Σε ορισμένες χώρες μπορεί κάτι τέτοιο να ισχύει, μπορεί να είναι αποτελεσματικό, αλλά σε άλλες χώρες όχι. Και ελπίζω η νέα, το νέο σώμα της Επιτροπής να μπορεί να δώσει μια πιο ικανοποιητική απάντηση εδώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αναφέροντα για την αναφορά αυτή. Πριν να εκλεγώ ως Ευρωβουλευτής, ε, ήμουνα επικεφαλής της Ευρωπαϊκής ε, Γραμματείας και είδα πώς λειτουργεί το σύστημα από το 2008 μέχρι πριν από δύο χρόνια. Και ο αναφέρον έχει απολύτως δίκιο. Και αν δεν κάνω λάθος, πριν από δυόμιση χρόνια υπήρξε μια ανακοίνωση από την Επιτροπή για Ε, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Πιλωτικό Σύστημα. Γιατί ορισμένα στοιχεία τα οποία διαπιστώθηκε δεν λειτουργούσαν καλά ε, και προκειμένου να υπάρξει μια μεγαλύτερη ευελιξία πριν ολοκληρωθεί η επίσημη ε, διαδικασία Ε, άρα λοιπόν ε, τελικά καταλήγουν ε, οι διαδικασίες αυτές, οι παραπομπές αυτές των χωρών μελών. Και χρειαζόμαστε ένα σύστημα το οποίο να δουλεύει. Εγώ προτείνω να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά ή να αποσταλεί στην Νομική Επιτροπή και επίσης να διαβιβαστεί στον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή όσον αφορά ειδικά την ε, λειτουργία αυτού του συστήματος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σαλίπα, έχετε, μπορείτε να κάνετε μόνο ένα... Ε, θέλω να σας κάνω το εξή σχόλιο. Ε, έχουμε... έχει γίνει αυτή, έχει διαβιβαστεί στην νομική επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ήδη είπατε ότι έχουμε μια γνωμοδότηση από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για την αναφορά αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αναφέροντα, αλλά πράγματι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων υπογράμμισε ότι το δικαστήριο διευκρινίζει ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση. Και επίσης η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σημαντικό να μειωθεί η εξουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών επί παραβάση θεωρούν ότι όλες οι διαδικασίες που έχουν στο σκοπό να τροποποιήσουν την ε, κυριαρχία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων προποθέτουν μια τροποποίηση των ευρωπαϊκών συνθήκων. Γι' αυτό από νομική άποψη πιστεύω ότι η κατάσταση είναι ξεκάθαρα. Αλλά βεβαίως συμφωνώ με τους συναδέλφους μια βελτίωση των διαδικασιών θα ήταν ε, κάτι το σημαντικό και βεβαίως θα είναι πρόσδεκτη από τους ε, πολίτες γιατί θα ξεκαθαρίσει το τοπίο ε, και θα διευκολυνθούν τα πράγματα για τους πολίτες. Αλλά δυστυχώς δεσμευόμαστε νομικά από τις συνθήκες και συνεπώς προτείνω να κλείσει η αναφορά αυτή. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω τους αναφέροντες. Κατά την άποψή μου, ο ρόλος της Επιτροπής, όπως ορίζεται από τις συνθήκες, είναι του θεματοφύλακα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ωστόσο, συχνά, πολύ συχνά, βλέπουμε η Επιτροπή δεν δρά αμερόληπτα. Συχνά δρά με διαφορετικό τρόπο. Αντίθετα, η Επιτροπή πρέπει να δρά με αμερόληπτο τρόπο προς, με στόχο την εξασφάλιση ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τα δικαιώματα των πολιτών που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εφαρμόζεται με ίδιο τρόπο παντού, ώστε να μην υπάρχει χώρος για διακρίσεις, αποφεύγοντας να δημιουργηθούν έτσι πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στην Ένωση. Όπως ξέρουμε ωστόσο, συχνά συμβαίνει αυτό. Τα παραδείγματα της αναφοράς είναι ξεκάθαρα. Υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες για, τα, ε, για τις συμβάσεις ε, περιορισμένου, περιορισμένης ε, διάρκειας από το 2013 και μετά. Κάθε μέρα ε, η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση ανοίγει την δυνατότητα, περιορίζει τη δυνατότητα προσλήψεων με επιχειρήματα δημοσιονομικού χαρακτήρα η Επιτροπή δεν λέει τίποτα γι' αυτά, ενώ θα μπορούσε να ε, αναλάβει δράση. Σε άλλες περιπτώσεις κατηγορεί τα κρατημέλη όταν προσπαθούν να δαπανίσουν χρήματα, τώρα κοιτάει από την άλλη μεριά. Αυτή η συζήτηση γίνεται μία εβδομάδα μετά την έγκριση από το Κοινοβούλιο ενός ψηφίσματος για την διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης που έχει μεγάλες φιλοδοξίες να φτιάξει ε, την εικόνα του μέλλοντος της Ευρώπης και ενδεχομένως την αναθεώρηση των συνθήκων. Πιστεύω εν ώψη αυτού να εκφράσουμε ως Κοινοβούλιο την ανάγκη να υπάρξουν σαφή κριτήρια για, την, για το πώς ξεκινούν οι διαδικασίες παραπομπές. Να αφαιρεθεί από την Επιτροπή το κυρίαρχο δικαίωμά της να αποφασίζει πότε θα παραπέμπει και ποιου, και ποια θα είναι προτερ, θέματα προτεραιότητας. Να μπει στο περιθώριο η λογική που είναι επικίνδυνη ότι υπάρχουν πολίτες που δικαιούνται προστασίες και πολίτες που δεν δικαιούνται. Κάτι που προέκυψε σε όλη την περίοδο Γιούνκερ. Στην τελευταία ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρει ότι η Επιτροπή θα διακρίνει τις περιπτώσεις με, την προστιθέμενη, με βάση την προστιθέμενη αξία που μία παραπομπή θα έχει και θα την κλείσει όταν, κλεί, όταν κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο από πολιτικής απόψεως. Άρα η Κομισιόν μιλάει για πολιτική ε, κρίση, όχι για την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις, όπως θα έπρεπε να δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαιοσύνη κάτω από τέτοιες συνθήκες. Ζητώ λοιπόν και κλείνω να μην ανοιχτεί η αναφορά για να μπορέσει το θέμα αυτό να μπει στις συζητήσεις για τις επόμενες φάσεις της μεταρρύθμισης των συνθήκων. Μια διαδικασία που τώρα ε, ξεκινά και να παραπεμφθεί στην Επιτροπή ΑΦΚΟ. Χρήσιμο είναι νομίζω. Να ζητήσουμε επίσης από την Επιτροπή μια ενημερωμένη πληροφόρηση για το θέμα αυτό. Να πω κι εγώ δύο λόγια. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ακούμε εδώ πολλά πράγματα. Η ευθύνη, η κύρια ευθύνη εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσία εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Commission has all possibilities to see in early stage of implementation. Η Επιτροπή έχει στόχο όχι να εφαρμόζει, αλλά να εξετάζει αν τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν. Η στρατηγική της Ένωσης που μας είχε απασχολήσει στο παρελθόν ε, για την αποφυγή των διακρίσεων έδειξε ότι πολλά κράτη είχαν ε, αποτύχει σε μια σειρά ε, δραστηριοτήτων υλοποίησης ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά η Κομισιόν έλεγε ότι δεν έχει χρόνο, δεν μπορεί να προλαβαίνει να ερμηνεύσει, την να, να μεταφράσει την εθνική νομοθεσία, να την καταλάβει κλπ. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν σαφές ότι δεν λάμβανε υπόψη την πραγματικότητα. Τι ζητάμε από την Επιτροπή. Δραστηριότητα, να είναι πιο ενεργή. Σήμερα για παράδειγμα. Ακούσαμε πολλές αναφορές για τα ζώα συνοδείας. Η Κομισιόν τι μας λέει. Δεν είναι αρμοδιότητα της Κομισιόν, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ιδέες όμως για το πώς θα γίνει αυτό αρμοδιότητα της Ένωσης δεν έχουμε. Είχαμε, α πούμε, την περίπτωση των ε, αναφερόντων από τη, Λιθουανία, από τη Λιθουανία. Δεν ξέρανε τι πρέπει να κάνουν για να έχει μια πραγματική επίδραση σε εθνικό επίπεδο ένας αναφέρον πρέπει να έχει χρήματα, δικηγόρους, ε, Αυτό θα το μπορούσαμε να το περάσουμε και στο scoreboard της Ένωσης. Στην Κύπρο μας είπε η αναφέρουσα θέλει έξι έως και 10 χρόνια μια υπόθεση για να περάσει όλο το δικαστικό σύστημα. Αυτά ήθελα να σας πω. Να τα λάβει η Κομισιόν αυτά υπόψη. Εδώ είστε. Μία πρόταση άκουσα μόνο, να μην ανοιχτεί η αναφορά. Και εσύ συμφωνείτε, ε, κύριε Άγιος Σαλίμπα. Yeah. So, no, no, I know. But we, we give two minutes to petitioner. Να δώσουμε βέβαια δύο λεπτά στον αναφέροντα. Αλλά μόνο αν μιλάει κανονικά, όχι τρέχοντας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμείς ε, δεν αναφερόμαστε σε διαδικασίες ε, παραβάση, σε ανούσια προβλήματα. Όταν ο Πάολο Βόλπε παρουσίασε την αναφορά, αναφερόταν σε διαδικασίες επί παραβάση που αφορούν διαρθρωτικά προβλήματα και όχι μόνο ε, σε ιταλικό πλαίσιο, αλλά σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Στις 31 Μαου του 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλειά του ενέκρινε το ψήφισμα κατά της επισφάλειας των εργασιακών σχέσεων. Ήδη από εκείνο το ψήφισμα καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ζητά να ε, παρακολουθεί πιο προσεκτικά το κοινοτικό δίκαιο. Το ψήφισμα αυτό γεννάται από την Επιτροπή Αναφορών. Εδώ δηλαδή γεννήθηκε. Και γεννήθηκε διότι δεκτήκατε τα αιτήματα των αναφερόντων και καταφέρατε ως Επιτροπή να τα φτάσετε στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και το Κοινοβούλιο αποφάσισε να περάσει ένα ψήφισμα το οποίο για την Ιταλία αλλά και για άλλα κράτη-μέλη ήταν πάρα πολύ σημαντικό και στην Ιταλία ένα μήνα μετά οδήγησε σε μια διαθεωτική μεταρρύθμιση των ε, συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Επομένως, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν μπορεί να τον υποκαταστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι συνεχείς καταγγελίες ε, των αναφερόντων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα και τελευταίο παράδειγμα. Σε απάντηση στο αίτημα να κλείσει η αναφορά στις 28 Νοεμβρίου του 2019, δηλαδή πριν από δύο μήνες περίπου, κάτι λιγότερο. Στο δικαστήριο συζητήθηκε μια πολύ σημαντική υπόθεση για το νομικό καθεστώς ε, του... Contesto il problema. Voi l'avete affrontato, voi l'avete portato in για ε, τους αμυστή δικαστικούς. Εσείς είστε αυτοί που θέσατε το θέμα στο Κοινοβούλιο. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε προστασία ενός πάρα πολύ ουσιαστικού ε, κομμάτος, ε, κομματιού της ε, Ιταλικής δικαιοσύνης που δεν προστατευόταν συμπεριλήφθηκε σε αυτό το ψήφισμα. Και μάλιστα ο δικαστής ε, της παραπομπής σε αυτή την περίπτωση πρότεινε να υπάρχει και ε, προσφυγή κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ρώτησε το δικαστήριο εάν μπορεί ο ίδιος ο Εθνικός Δικαστής να ενεργοποιήσει μία δράση για αποζημίωση ε, στην Ιταλία ενώπιον του Εθνικού Δικαστή για μη τήρηση της οδηγίας και των συνθήκων από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το να κλείσει λοιπόν αυτή η υπόθεση σημαίνει ότι θα ανοίξουμε μια υπόθεση γιατί κάποιο ε, θα καταγγείλει το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκλεισε τη διαδικασία επί παραβάση, διαπιστώνει ότι υπάρχει μια διορθωτική κρίση και παρόλα αυτά δεν έκανε τίποτα. Το έκανε με του αμυστή δικαστικού, το έκανε λοιπόν και με τι ε, ε, συμβάσει ορισμένου χρόνου. Εσεί παρεμβήκατε και θα πρέπει να παρέμβετε και τώρα ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εποπτεύει σωστά και εγκαίρως ε, την εφαρμογή των συνθήκων και ίσως και προτείνοντας και αλλαγή των συνθήκων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ντεμικέλε. Και τώρα θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε και να αποφασίσουμε όλοι όσοι πήραν το λόγο πρότειναν ε, να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. και να δούμε τι θα γίνει. Και πώς θα λάβει υπόψη της το αίτημα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο δραστήρια για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας από πλευράς κρατών μελών. Η κυρία Εύη, παρακαλώ. Μπορούμε να το στείλουμε και στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για να γνωμοδοτήσει. Έχουμε ήδη γνωμοδότηση από τη Γιούρη. Να το στείλουμε και στην ΑΦΚΟ. Τι λένε οι συνάδελφοι. Ο κύριος Βίντσε, ο κύριος Σαλίμπα. Ναι. Ε, εντάξει, θα το στείλουμε στην ΑΦΚΟ λοιπόν την αναφορά. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι πλέον ε, εξαντλήσαμε την ημερήσια διάταξη. Θα τα πούμε στην επόμενη συνεδρίαση, η οποία θα γίνει 20... Κάπου εδώ πρέπει να είναι.